gentlemen. Um, Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Κάριν Κόλμαν είμαι, Ιρλανδή δημοσιογράφος και θα διευθύνω τις επόμενες ε, δύο συζητήσεις ε, και σφαρσιάζω τους καλεσμένους μας, τον κύριο Ζαν Κλοντ Τρισέ, τον οποίον φαντάζομαι ότι ξέρετε, πρώην ε, διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, από το 2003 μέχρι το 2011 και όπως ξέρετε τα τελευταία χρονάκια ε, της θητείας του είχε να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα είναι πρόεδρος του ΔΣ του Μπρούγκελ, ε, της ομάδας των Τριάκοντα και ευρωπαϊκός πρόεδρος της Τριμερούς Επιτροπής και κάποια άλλα αξιώματα βεβαίως κατέχει αλλά οπωσδήποτε τα βασικά είναι αυτά. Να σας πω τώρα τι θα γίνει. Θα ήθελα να μας πει ο κύριος Τρισέ πώς βλέπει τα πράγματα ως πρώην διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πώς βλέπει την κατάσταση, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οικονομικό και ξέρω πως πολλοί ε, από εσάς ε, θα θέλετε να θέσετε ερωτήσεις και ευχαρίστως θα απαντήσει. Κύριε Τρισέ, σας καλωσορίζω ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο πρωτοήρθατε νομίζω το 2003, όταν πρωτογίνατε διοικητής. Σας ευχαριστώ. Κάριν. Μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ. Αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι στα γαλλικά. είμαι ιδιαίτερα συγκινημένο που είμαι πάλι στις αίθουσες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από τόσα χρόνια. Γιατί όταν ήμουν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχω, είχα έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνω από 40 φορές. Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έβρισκε τη μεγαλύτερη αμεσότητα, τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη παρά τις διαφορετικές απόψεις που επικρατούσαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από ιστορική έποψη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησαν στην αρχή ξεκίνησε η εντολή μου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στον Νοέμβριο του 2003 διορίστηκα επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας. Εξήγησα στους βουλευτές πόσο σημαντικό ήταν να μπορέσουμε να σεβαστούμε μέχρι κεραία στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό ένα πλαίσιο για τον προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είχαμε το ενιαίο νόμισμα αλλά δεν είχαμε καμία κοινή πολιτική σε επίπεδο δημοσιονομικών θεμάτων. Επομένως έπρεπε να σεβαστούμε το πλαίσιο αυτό το οποίο ήταν είχε θεσπιστεί για την ζώνη του ευρώ. Είδαμε μετά ποιες ήταν οι συνέπειες οι οποίες προέγυψαν. Το Δεκέμβριο του 2003 ήδη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχα τονίσει την ανάγκη σεβασμού αυτού του πλαισίου. Όταν ξεκίνησε όμως η κρίση από το 2007, εγώ είχα την ευκαιρία να μεταφέρω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις απόψεις μου για την κρίση των ομολόγων subprime, την κατάρρευση της Lehman Brothers και την οικονομική κρίση που ακολούθησε. Όταν η χρηματοπιστωτική κρίση από κρίση ομολόγων πέρασε σε κρίση κρατικού χρέους και μετά σε οικονομική κρίση. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που είμαι εδώ πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, επειδή μιλήσατε για την ευρωπαϊκή κρίση, κύριε Τρισέ. Τώρα, το 2014, δυόμιση χρόνια μετά την αποχώρησή σας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ίσως ήταν ένα δύσκολο χρονικό διάστημα και για σας, πώς θα περιγράφατε την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο. Θα ήθελα να σας δώσω την δική μου εικόνα για την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Είχαμε την κρίση των ομολόγων δεύτερης ποιότητα, τον Αύγουστο του 2007, τα λεγόμενα subprime. Αν θυμάστε, στις 9 Αυγούστου 2008 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να παράσχει απεριόριστη ρευστότητα σε όλες τις αντισυμβαλόμενες τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μας ζητήσαν 95 δισεκατομμύρια ευρώ. <clears throat> Ήταν η πρώτη λοιπόν δράση μας τον καιρό της κρίσης. Ήταν στη φάση που ήταν ακόμα τα ομόλογα subprimes. Μετά κατέρευσε η επενδυτική τράπεζα Lehman Brothers που οδήγησε σε μια πολύ σοβαρή απειλή για κατάρρευση του συνολικού χρηματοπιστωτικού συστήματος ήταν μια δραματική κατάσταση και αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπως και κάποιες άλλες τράπεζες όπως η Federal Reserve στις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν είχαμε δράσει με ένα ταχύ και τολμηρό τρόπο τότε θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε την πιο σοβαρή ύφεση μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όχι την ε, χειρότερη ύφεση, αλλά την χειρότερη βαθιά οικονομική κρίση. Ήταν τόσο απειλητικά τα πράγματα όπως τα έβλεπα εγώ. Και μετά είχαμε ένα τρίτο στοιχείο σε αυτή την αλληλουχία γεγονότων, όταν τροποποιήθηκε η κρίση από τον ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα σε κρίση του δημόσιου χρηματοπιστωτικού τομέα. Όταν η κρίση των subprimes και της Lehman Brothers έγινε κρίση κρατικού χρέους. Η μετάβαση λοιπόν από το δεύτερο επεισόδιο στο τρίτο επεισόδιο της, κρίτη, της κρίσης, η κίνδυνη για τα κρατικά ομόλογα, ήταν τότε που σε συντονισμό με τον Μπεν Μπερνάνκε χρειάστηκε να δράσουμε. Μου είπε στη Βασιλεία ο Μπεν Μπερνάκη, κοίτα Ζαν Κλοντ, σειρά σου είναι τώρα. Το επίκεντρο της κρίσης δεν είναι πια στις ΗΠΑ, αλλά έχει περάσει τον Ατλαντικό. Εμείς βρεθήκαμε στο μάτι του κυκλώνα μετά από την κατάρρευση της ε, Lehman Brothers. Τώρα όμως το επίκεντρο του επόμενου, της επόμενης κρίσης βρίσκεται στην Ευρώπη. Είναι η δικιά σας σειρά να κάνετε κάτι. Είχε δίκιο λοιπόν ο Μπεν. Ήταν μια πολύ καλή εικόνα της κατάστασης και εμείς χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε το τρίτο στάδιο της κρίσης μετά από την αντιμετώπιση των προηγουμένων εκδηλώσεων της κρίσης. Μπορώ να πω και περισσότερα, αν θέλετε. Ε, συναρπαστικό, γιατί σπάνια μπορούμε να μαθαίνουμε το πώς λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις. Πώς είχε η κατάσταση τις μέρες εκείνες όταν έπρεπε να λάβετε πολύ δύσκολες και γρήγορες αποφάσεις που θα επηρέαζαν εκατομμύρια ανθρώπους. Υπάρχουν δύο διαστάσεις. Η μία είναι να αντιληφθούμε το γιατί ήμασταν το επίκεντρο της παγκόσμιας ε, κρίσης όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα. Ποιες ήταν οι αδυναμίες ε, που εξηγούν το γιατί ήμασταν το επίκεντρο και Ακριβώς γιατί πήγε η σειρά Bear Stearns, Freddie Mac and Fannie Mae, Lehman Brothers, AIG που αποκαλύπτει τις ε, αδυναμίες του στήματος της ΕΠΑ. Πρώτα απ' όλα ποιες ήταν οι αδυναμίες, ε, γιατί ήμασταν το επίκεντρο της ε, κρίσης και ποιες αποφάσεις έπρεπε να λάβουμε για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Μια ανάγνωση είναι πως αντιλαμβανόσασταν, αν μου επιτρέπετε, την κατάσταση μεταξύς, μεταξύ ε, Κεντρικής Τράπεζας ε, του Εκτελεστικού Κλάδου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Είναι πάρα πολλές οι διαστάσεις. Ξέρω πως θα γίνουν και ερωτήσεις. Μπορείτε λοιπόν να με ρωτήσετε για όλα αυτά, αλλά για να συνοψίσω θα έλεγα πως για εμάς ήταν λυπηρό το να βλέπουμε ότι ήμασταν το επίκεντρο της ε, κρίσης και θα σας δώσω μόνο τίτλους αν θέλετε και μετά μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις για τους ε, έξι λόγους για τους οποίους κατά την άποψή μου ε, είχαμε το θλιβερό προνόμιο να είμαστε το επίκεντρο της κρίσης γιατί ήταν πάλι τμήμα της Ευρωζώνης αυτό το οποίο είχε τις μεγάλες δυσκολίες όχι ολόκληρη η Ευρωζώνη πρώτα απ' όλα δεν σεβαστήκαμε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, το ανέφερα, παρά το ότι βεβαίως ήταν προφανές ότι αναλαμβάναμε κίνδυνο. Δεύτερον, δεν επιτηρούσαμε τους, ε, αν, τους δείκτες ανταγωνιστικότητας, τις εξωτερικές ανισορροπίες που καταδείκνυαν την απώλεια ανταγωνιστικότητας μεταξύ των οποίων το μοναδιαίο κόστος εργασίας στις διάφορες χώρες. Πρέπει να πω πως η τράπεζα από το 2005 έβγαζε αυτούς τους δείκτες ανταγωνιστικότητας, ε, τους έδινε σε όλες τις κυβερνήσεις κάθε μήνα για να ε, γνωρίζουν ε, τις διαφορές που συσσωρεύονταν στην Ευρωζώνη. Τρίτον, δεν είχαμε τραπεζική ένωση και στην κρίση φάνηκε πως η σχέση μεταξύ φερεγγιότητας των κρατών και φερεγγιότητας των τραπεζών ήταν πάρα πολύ στενή, έτσι ώστε στην Ευρωζώνη είχαμε αφενός φαύλους κύκλους, αλλά και κάποιους θετικούς, αν θέλετε, ενάρετους, όπως λέμε, κύκλους μεταξύ της κρατών και τραπεζών. Αυτό το λάστο το έκαναν όλες οι χώρες. Η ε, και το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά στην Ευρωζώνη υπήρχε ακριβώς η διαφορά μεταξύ αυτών οι οποίοι πήγαιναν πάρα πολύ καλά και αυτών οι οποίοι είχαν βυθιστεί στην κρίση. Τέταρτος λόγος, δεν υπήρχαν εργαλεία εκ των προτέρων για να αντιμετωπίσουμε τη δραματική κρίση, οπότε έπρεπε να εφεύρουμε τους ε, μηχανισμούς, ε, το Ταμείο και το Μηχανισμό Μετασταθερότητας. Αυτοί είναι οι τέσσερις λόγοι. Αυτοί είναι συγκεκριμένοι και αφορούν ειδικά την ε, Ευρωζώνη. Και μετά υπάρχουν άλλοι δύο ε, λόγοι που ισχύουν και για τα 28 κράτη-μέλη της Ένωσης. Ε, ο πρώτος είναι πως δεν έχουμε επιτύχει ενιαία αγορά. Είναι λυπηρό για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ιδιαίτερα για την Ευρωζώνη, επειδή η Ευρωζώνη χρειάζεται πολύ ευέλικτη η οικονομία με ενιαία αγορά και τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό δεν εφαρμόστηκε πλήρως δεν εφαρμόστηκαν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πρόγραμμα της Λισαβόνας ε, το πρόγραμμα του 2020 κατά το οποίο είναι και πάλι πρόβλημα και για τους 28 αλλά ιδιαίτερος για την Ευρωζώνη όσον αφορά ειδικά την ευελιξία των οικονομιών και την δυνατότητά τους να αντιμετωπίσουν την κρίση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ακριβώς τις ανισορροπίες με το σωστό τρόπο. Υπάρχουν λοιπόν οι έξι λόγοι, τίτλοι κεφαλαίων όπως σας είπα, οπότε δεν λάβαμε με βάση αυτά κάποιες αποφάσεις. Πρώτα απ' όλα ενισχύθηκε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξη. Υπάρχει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και σημαντικό η αναστροφή του βάρους της αποδείξεως. Δηλαδή, εάν το Συμβούλιο θέλει να κάνει κάτι αντίθετο από την πρόταση της Κομισιόν, πρέπει να έχει πλειοψηφία για να ανατρέψει την απόφαση της Κομισιόν. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει αντιστροφή του βάρους αποδείξεως και πραγματικά ε, οφείλω να επενέσω το κοινοβούλιο το οποίο ακριβώς ε, ζήτησε αυτό το πράγμα. Κατόπιν τώρα επιτηρούμε τους ε, δείκτες ε, της ανταγωνιστικότητας είναι η λεγόμενη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών και θα ήθελα να συγκρατήσετε το εξής. Η διαδικασία αυτή μακροοικονομικών ανισορροπιών είναι κατά την άποψή μου εξίσου σημαντική με το σύμφωνο ε, σταθερότητας και ανάπτυξης ε, γιατί κάποιες χώρες είχαν προβλήματα επειδή δεν σεβάστηκαν το σύμφωνο άλλες ε, βρίσκονταν σε μία φούσκα και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ότι έχαναν ανταγωνιστικότητα και ότι θα ήταν πολύ ευάλωτες. Οπότε θα χρειαζόμαστε και τα δύο. Και σε μία νομισματική ε, ένωση πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη το ότι πέρα από ονομαστική πρέπει να, πέρα από ονομαστική πρέπει να παραμένει και πραγματική ενιαία ζώνη. Να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις και αυτό σημαίνει πως πρέπει να παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά τους δείκτες ανταγωνιστικότητας, το μοναδιαίο κόστος εργασίας και έτσι ώστε οι ονομαστικοί δείκτες να μην αποκλίνουν πολύ από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτά είναι, αυτές είναι οι δύο πρώτε διορθώσει που έγιναν για τι αδυναμίες. Για την τρίτη αδυναμία ξέρετε πω έχουμε τώρα την Τραπεζική Ένωση, κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο πριν από την κρίση και είχε καθυστερήσει βεβαίω ε, ήδη, τώρα εφαρμόζεται όπω γνωρίζετε, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό, αλλά νομίζω πω ε, κάτι το πάρα πολύ σημαντικό είναι η δημιουργία, όπω είπαμε, τη ε, τραπεζική Ένωση και της διαδικασίας της ε, παρακολούθησης αυτής των δικτών που είναι πάρα πολύ σημαντικά της οικονομικής διακυβέρνησης και δημιουργήθηκε και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, δεν θα επιμείνω σε αυτό. Εγώ οπωσδήποτε θα, θα ζητούσα να επιτευχθεί η κοινή αγορά και η στόχη του προγράμματος 2020 γιατί έχουν ουσιαστική σημασία για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη όπως είπα. Οπότε, εδώ είμαστε λοιπόν μετά από την χειρότερη κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο και μετά που θα μπορούσε ε, να είναι και η χειρότερη κρίση από τον Πρώτο Παγκόσμιο όπως ήδη εξήγησα και αν μου επιτρέπετε Καρίν θα ολοκληρώσω εκεί θα τονίσω ε, λίγο παραδόξως ίσως τη στιγμή αυτή την οποία μιλάμε την αντοχή της Ευρώπης και της Ευρωζώνης. Γιατί θα θυμάστε πως στην αρχή υπήρχε η αίσθηση εκτός και ίσως και εντός Ευρώπης πως το ευρώ θα εξαφανιστεί ως νόμισμα και δεν είναι δυνατόν να αντέξει σε μια τέτοια κρίση, τη χειρότερη κρίση από το Δεύτερο Παγκόσμιο και θα αποσυνδεθεί η Ευρωζώνη και δεν ε, μπορεί να είναι τόσο τολμηρή και τόσο θρασής ώστε να αντέξει το ευρώ. Τι να πω τώρα λοιπόν. Πρώτον, το ευρώ ως νόμισμα ήταν πάντα αξιόπιστο καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης όπως ίσως ξέρετε είναι πάνω από την αρχή του ισοτιμία με το αμερικανικό δολάριο καθ' όλη τη διάρκεια της ε, κρίσης από την εποχή της ε, Lehman Brothers. Μπορεί να προξενεί έκπληξη το βασικό πρόβλημα του ευρώ, όπως ξέρετε, ήταν ότι σκεφτόμασταν πως είναι πολύ δυνατό ε, παράδοξο για, μια, για ένα νόμισμα το οποίο υποτίθεται πως είναι ασθενές. Δεύτερον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, Ήμασταν 15 μέλη της Ευρωζώνης ε, τη στιγμή της Lehman Brothers. Οι 15 εξακολουθούν να είναι μέσα στο ευρώ σήμερα μετά από όλα αυτά την πολύ δύσκολη περίοδο. 2009 και είμαστε τώρα στο 2014. Οι 15 χώρες, οι 15 δημοκρατίες αποφάσισαν να μείνουν εντός και αυτοί που είχαν προβλήματα υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Και ε, όσοι δεν είχαν θυχτεί αποφάσισαν να βοηθήσουν ακόμα και αν δεν ήταν εύκολο και το αντιλαμβάνεστε όλοι το γιατί. Επιπλέον τρεις νέες χώρες μπήκανε τη στιγμή της κρίσης 15 ε, τη στιγμή της Λίμαν 18 χώρες σήμερα Τρεις χώρες εντάχθηκαν, όπως ξέρετε, η Σλοβακία, η Λετωνία Η Σλοβενία είχε μπει πριν. Και η Εστονία, ναι. Και η Λιθουανία μπορεί να μπει το... τον επόμενο Ιανουάριο. Δεν μετράω τη Λιθουανία. Τρεις χώρες λοιπόν ακόμα. Κάτι λοιπόν το οποίο δείχνει πως ε, η αντοχή του ευρωπαϊκού οικοδομήματος ε, οπωσδήποτε είναι μεγαλύτερη από ό,τι φανταζόμασταν ε, εκ των προτέρων. Δεν συμπεραίνω πως όλα πηγαίνουν μια χαρά. Όπως ξέρετε ο εφησυχασμός είναι το χειρότερο δυνατόν. Έχουμε πολλά να κάνουμε, αλλά εγώ αντιλαμβάνω πως ε, το ιστορικό αυτό έργο, αυτό η οικοδόμηση της ε, Ευρώπης ε, και η σημασία του και η δύναμη του ίσως να μην γίνεται πάρα πολύ καλά αντιληπτή απ' έξω γιατί είναι πολύ τολμηρό πράγματι και δεν μπορεί κανείς απ' έξω να αντιληφθεί το τι σημαίνει αλλά είχαμε και τα τεστ και τα οποία περάσαμε και αυτά τα οποία σας είπα είναι αντικειμενικά γεγονότα. Είμαστε 18 χώρες αυτή τη στιγμή, καμία χώρα δεν έχει φύγει και βεβαίως το νόμισμά μας ήταν αξιόπιστο καθόλου. αυτή τη διάρκεια. Σημαντικό. Ακόμα και αν γεγονός είναι πως το βασικό πρόβλημα είναι πως είναι πολύ ισχυρό. Και πρέπει να το δούμε και αυτό βεβαίως. Μία τελευταία δες προς τον κύριο Τρισέ πριν δοθεί οι σχετικοί δημοσιογράφους γιατί βέβαια πάρα πολλοί έχουν χτυπηθεί από αυτά τα σκληρά μέτρα στα οποία επέμεινε η ΕΚΤ ε, ήταν το θέμα του πληθωρισμού και σε κάποιες χώρες όπως στην Ελλάδα είχαμε πει ότι εάν δεν γίνει κάτι θα βγουν από την Ευρωζώνη. Όμως ε, αυτή τη στιγμή αυτό που κληροδοτήθηκε είναι μια μακροπρόθεσμη φτώχεια και τελικά ότι από όλα αυτά ωφελήθηκαν οι πλούσιοι Γερμανοί και οι άλλοι και οι άλλοι πλούσιοι της Ευρώπης. Τρισέ. Πρώτα πρώτα όπως σας προανέφερα. Η Καπατάφ είπε ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστό πάνω απ' όλα το σύμφωνο σταθερότητας. Εάν είχε γίνει σεβαστό, εάν είχε τηρηθεί στις ε, χώρες όλες αυτές, δεν θα υπήρχαν αυτά όλα τα σοβαρά προβλήματα ούτε στην Ελλάδα. Οπότε το να πει κανεί ότι ευθύνεται η ΕΚΤ για αυτά τα προβλήματα καθιονδήποτε τρόπο, ε, τότε αυτό αντιβαίνει 100% στην ε, αλήθεια, στην πραγματικότητα. Γιατί η πραγματικότητα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη για όλε τι κυβερνήσει. Τώρα, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, το καμπανάκι του κινδύνου ξεκίνησε πολύ πριν ξεκινήσει η κρίση. Πέντε χρόνια πριν έχουμε την κρίση του κρατικού δημοσίου χρέους. Ήταν ξεκάθαρο ότι υπάρχει πρόβλημα από τότε. Και κάποια συγκεκριμένη χώρα, πώς να πω που ήταν η πιο αδύναμη, είχε 15% του ΑΕΠ έλλειμμα τρέχουσών συναλλαγών. Γνωστό ε, αυτό το ποσοστό. Και έτσι φτάσαμε στην τραγωδία. και όχι μόνο από το γεγονό ότι θα έπρεπε να έχει γίνει διορθωτική κίνηση. Και από ό,τι γνωρίζω είναι ότι η χώρα η οποία δεν έχει κανένα πρόβλημα στην κρίση, τέλο πάντων ε, οι χώρε οι οποίε είχαν τα πιο λίγα προβλήματα είναι οι χώρε οι οποίε ήταν πριν προσεκτικέ, φρόνιμε. Και αυτέ και αμύθηκαν. Και γι' αυτό και είχαμε αυτή την ε, εξέλιξη, ε, διαφορά του μοναδίου 26 των χρόνων αυτών που είναι γιγαντιαία. Βεβαίω και υπήρχε δυσκολία προσαρμογή, αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφευθεί είναι το να δημιουργηθούν οι ανισορροπίες οπότε και θα έπρεπε να γίνει κατόπιν υποχρεωτικά αυτή η διόρθωση η προσαρμογή και γι' αυτό και θα πρέπει να εξηγηθεί το ότι στην συγκυρία αυτή τότε ήταν όλα εύκολα εύκολη χρηματοδότηση παρά τα καμπανάκια κινδύνου Οπότε ξεκίνησε έτσι το σπιράλ αυτό, η αντίστοφη μέτρηση για το χρέος. Βεβαίως και είχαμε και αντίκτυπο, είχαμε και συνέπειες από την Αμερικανική κρίση. Οπότε πια σταυρώσαμε τα χέρια, όλοι λέγανε δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η χρηματοδότηση του χρέους σας. Καθίστε και διορθώστε ο καθένας το δικό του έλλειμμα και επιστρέψτε σε μια ισοσκελισμένη κατάσταση. Επομένως, όλα αυτά μπορεί να τα κάνετε με τρόπο εντυπωσιακό ε, ή να το κάνετε σε αυτή την κλίμακα ή να το κάνετε αν όχι με τους ε, Ευρωπαίους φίλους να το κάνετε με κάποιους από την παγκόσμια σκηνή. Βεβαίως και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βεβαίως και είχαμε στο 15% οπότε και τότε θα έπρεπε κανείς να επιστρέψει κοντά στο μηδέν πλεόνασμα. Γιατί δεν υπήρχε δεκάρα για να χρηματοδοτηθεί τίποτε. Με, αφού υπήρχε, είχαμε φτάσει στο, στο πλήν 15%. Αυτή ήταν η πικρή αλήθεια. Άρα και θα έπρεπε επομένω να εφαρμοστεί κατά γράμμα αυτή η νέα διακυβέρνηση που προβλεπόταν εν εν θερμό. Η Τραπεζική Ένωση, ε, το MIP που προαναφέραμε και όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν όσο γίνεται πιο ανοιχτά, πιο αυστηρά. Πολύ σημαντική για μένα αυτή η νέα διακυβέρνηση, αλλά όμως πέραν αυτών θα πρέπει να προγραμματιστούμε για το μέλλον. Και ο ίδιος έχω υποβάλει προτάσεις όσον αφορά στο μέλλον. Ε, εάν ενδιαφέρεστε να σας αναλύσω το τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον και δεν εννοώ εδώ και τώρα, αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον γιατί θα πρέπει να έχει περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έρχονται τώρα οι ευρωεκλογέ. Και θα πρέπει να υπάρχει δημοκρατική υποχρέωση λογοδοσίας ε, από πλευρά των Ευρωπαϊκών Θεσμών Οργάνων και αυτό θα πρέπει να γίνεται προ το Κοινοβούλιο. Τώρα δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση λογοδοσίας σε αυτό το όλο το, το, στερέωμα των θεσμικών οργάνων της Ευρώπης. Η Πρόεδρος. Ε, ευχαριστούμε και τώρα από το Ακροατήριο. Πρώτα-πρώτα οι κύριοι πίσω-πίσω στην αίθουσα, οπότε παρακαλώ πρώτα-πρώτα να πείτε το όνομά σας και από το έντυπο ή κανάλι από το οποίο προέρχεστε. Στέφαν. Στέφαν Σευρυπίδου, από μια Κυπριακή εφημερίδα. Είμαι μία από τη... Η Κύπρος είναι μία από τις 15 δημοκρατικές χώρες που είναι στο ευρώ. Μιλήσατε για το σύμφωνο ανάπτυξης και σταθερότητα ότι είναι ένα πρόβλημα για πολλές χώρες. Θα ήθελα να σχολιάσετε το, την περίπτωση της Κύπρου, όπου οι τράπεζες ήταν αυτές οι οποίες είχαν υπερθερμανθεί ουσιαστικά, αλλά είχαν και μεγάλη έκθεση σε κρατικά ομόλογα και αυτό οδήγησε σε μια κατάσταση που η κυβέρνηση δεν μπορούσε να τις υποστηρίξει. Αυτό οδήγησε στο πρώτο bail-in, το οποίο ορισμένοι θεωρούν ότι ήταν απλώς αρπαγή των καταθέσεων των καταθετών. Και αντίθετα από αυτά που λέγανε οι γερμανικές εφημερίδες, δεν ήταν όλοι οι Ρώσοι ολιγάρχες, πολλοί Κύπροι έχασαν τα λεφτά τους. Θα ήθελα λοιπόν τα σχόλιά σας, γιατί αυτό νομίζω ότι αλλάζει την αντιμετώπιση ότι το σύμφωνο σταθερότητα ήταν το μόνο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ σύντομα. Δεν θέλω να σταθώ πάρα πολύ σε ένα μονάχα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να εξηγήσει λοιπόν η μη τήρησή του πολλά από τα προβλήματα, αλλά και η Τραπεζική Ένωση ήταν ένα σημαντικό στοιχείο και οι κανόνες διακυβέρνησης γενικά σε επίπεδο προϋπολογισμού και σε επίπεδο χρηματοπιστωτικό. Η περίπτωση της Κύπρου ήταν πραγματικά όλος ιδιαίτερη, γιατί είναι μικρό το ΑΕΠ της χώρας αυτής. Το μέγεθος του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι γιγάντιο και η χρηματοδότηση που πήρε η Κύπρος από την υπόλοιπη Ευρώπη ήταν πολύ μεγάλη ως ποσοστό του ΑΕΠ της σας τα αναφέρω όλα αυτά, αν δεν τα έχετε αυτά υπόψη σας, τότε δεν κατανοείτε πλήρως τις αποφάσεις που πήραμε. Η κυβέρνηση της ε, Κύπρου ως ε, τελική καταφύγη, γιατί τελικά όλες αυτές οι αποφάσεις ελήφθησαν από την Κύπρο. Και η κυβέρνηση λοιπόν και η Κυπριακή Βουλή με την υποστήριξη της υπόλοιπης Ευρώπης πήρε αυτές τις αποφάσεις. Ήταν μια τελείως ιδιαίτερη περίπτωση, μοναδική περίπτωση. Μάλιστα, ο κύριος εδώ μπροστά και εσείς πίσω, ο κύριος με το ροζ που κάμισο. Ή χαίρομαι που βλέπετε το χρώμα του πουκαμίσου μου. Κύριε Τρίσε, η Δανία από την οποία προέρχομαι δεν είναι τμήμα του, της ζώνης του ευρώ. Τα, νομίσματά μας, τα χαρτονομίσματά μας λοιπόν δεν έχουν το ίδιο χρώμα με το ευρώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όταν κάθεστε εσείς, όταν καθόσετε στο γραφείο σας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι χώρες αυτές που δεν ήταν στη ζώνη του ευρώ, όπως ήταν η Μεγάλη Βρετανία και η Δανία, πώς αντιμετωπίζετε. Έχετε απόλυτο δίκιο όταν κοίταζα τις 15 χώρες της ζώνης του ευρώ, υπολόγιζε και την Δανία ότι ήταν μία από αυτές. Γιατί όπως ξέρετε η Δανία παρακολουθεί τον πυρήνα του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος από πολύ κοντά. Είναι λοιπόν τμήμα της ευθύνη μας να είμαστε σε στενή επαφή με την Κεντρική Τράπεζα της ε, Δανίας και ήταν πάρα πολύ στενές και φιλικές οι σχέσεις μας. Η Δανία λοιπόν, όπως είπατε, είναι de facto τμήμα της ζώνης του ευρώ. Αν πάρω τώρα τις χώρες που ήταν ε, γενικά εκτός της ζώνης του ευρώ, πρέπει να πω ότι όλες μου οι επαφές κατά τη διάρκεια της κρίσης, της πιο δύσκολης εποχής της κρίσης, μετά από την κατάρρευση των ε, της ε, Lehman Brothers και μετά από τις πρώτες ε, απαρχές της κρίσης τον Αύγουστο του 2007 είχαμε μια πολύ στενή σχέση με τις χώρες αυτές και όλοι οι συναδελφοί μου, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια <clears throat> πάντα ζητούσαμε η ζώνη του ευρώ να εξασφαλίσει την κατάλληλη σταθερότητα για να εξασφαλίσει τη γενική σταθερότητα και ευμάρεια. Δεν υπήρξε καμία λοιπόν διαφορά απόψεων σε σχέση με τον ουσιαστικό στόχο που ήταν η διατήρηση της σταθερότητας <clears throat> και η σωστή λειτουργία της ε, ζώνης του ευρώ, γιατί αν δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα είχαμε επιπτώσεις για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι χώρες λοιπόν που δεν ήταν στη ζώνη του ευρώ θα είχαν επιπτώσεις να αντιμετωπίσουν. Πίσω κάποιος κύριος ήταν και εσείς εδώ τώρα. Ο κύριος πίσω παρακαλώ. Είδα το χέρι σας να σηκώνετε. Από το Λουξεμβούργο. Για τη μεγαλύτερη εφημερίδα του Λουξεμβούργου. Το ερώτημά μου είναι, κύριε Τρισέ, είσαστε σίγουρος ότι έχει ξεπεραστεί η ευρωπαϊκή κρίση και είμαστε ασφαλείς τώρα. Γιατί η Ελλάδα και η Πορτογαλία και η Κύπρος είναι σχετικά μικρές χώρες. Τι θα γίνει όμως αν η Γαλλία ή η Ιταλία αντιμετωπίσουν πρόβλημα κρατικού χρέους. Ο Φρανσουάς Μπό, ένας Γάλλος πολιτικός επιστήμονας, δημοσίευσε ένα βιβλίο που ζητάει μια οργανωμένη διάλυση της Ευρωζώνης. Τι θα απαντούσατε σε αυτή την έκκληση. Να σας πω ότι διαφωνώ πλήρως με τον Φρανσουά Εσμπό όταν μέσα στην κρίση όλες οι χώρες όλες οι δημοκρατικές αυτές χώρες χωρίς καμία εξαίρεση πρέπει να αποφασίσουν αν θα μείνουν ε, στην ζώνη του ευρώ ή όχι είπαν όλες ότι θέλουμε να διατηρήσουμε την ακαιρεότητα της ζώνης του ευρώ, ακόμα και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ανεξάρτητα από το ιστορικό εγχείρημα το οποίο διακυβευόταν που είναι πολύ σημαντικό υπήρχαν και άλλοι πολλοί λόγοι για τους οποίους θα ήταν πραγματικά δραματικό για οποιαδήποτε χώρα να βγει από τη ζώνη του ευρώ. Όταν λέω οποιαδήποτε χώρα μεγάλη ή μικρή. Ακόμα και οι χώρες που είχαν προβλήματα και αυτές που δεν είχαν προβλήματα. Το δεύτερο σας ερώτημα. Το, το απάντησα το πρώτο σας ερώτημα. Αν έχουμε ξεπεράσει την κρίση. Αν δούμε τον υπόλοιπο κόσμο, όταν είμαστε στο Τόκιο, στη Σανγκάη, στη Σιγκαπούρη, στο Χονγκ Κόνγκ, στη Νέα Υόρκη ή και το Λονδίνο, βλέπω σημαντική αλλαγή σε σχέση με τις ε, διαγνώσεις που διατυπώνται για τη ζώνη του ευρώ. Πριν από μερικά χρόνια Λέγανε όλοι, μα θα καταρρεύσει σίγουρα, σίγουρα θα καταρρεύσει, σίγουρα θα εξανεμιστεί η ζώνη του ευρώ, θα φύγουν χώρες από την ζώνη του ευρώ, δεν θα μπορέσει να διατηρηθεί αυτή η ιδέα. Τώρα βλέπω ακριβώς το αντίθετο, όπως είπατε και ο ίδιος. Μπορούμε να δούμε πραγματιστικά και αν ήμουν επενδυτής ή αποταμιευτής σε παγκόσμιο επίπεδο θα έλεγα ότι και αυτοί κατάφεραν να η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να επιβιώσει, θα έπρεπε σαν επενδυτές αποταμιευτές να καταλάβουμε ότι έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας το επιβεβαίωσε αυτό η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, ακόμα και η Ελλάδα. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω από αυτά που λέτε είναι το εξή. Και σα το λέω και γιατί είναι και η προσωπική μου θέση. Ότι όλε αυτέ οι χώρε έκαναν τι απαραίτητε προσαρμογέ. Όλε οι χώρε οι οποίε βρέθηκαν σε μεγάλη ανισορροπία σε ό,τι αφορά ιδίω το ισοζύγιο τρέχουσών συναλλαγών που ήταν μείον 8,5% κατά μεσονόρο για τις πέντε χώρες οι οποίες υπέστησαν μεγάλη πίεση το 2008-2009 τώρα έχουν πλεονασματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνολικά. Έγινε λοιπόν μια πολύ σημαντική προσαρμογή. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό στοιχείο, δεν είναι υποκειμενικό. Δεύτερον, η νέα μορφή διακυβέρνηση που ανέφερα προηγουμένω υπάρχει. Ενισχύθηκε το σχέδιο ε, σταθερότητας και ανάπτυξης, το σύστημα εποπτείας για τα νομισματικά θέματα και η Τραπεζική Ένωση. Επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο ισχυρή και έχουμε ένα νέο σύστημα λοιπόν διακυβέρνησης που εδρεώθηκε το 2010 και το 2011. Τέλος, όλες οι δημοκρατίες, σας υπενθυμίζω, είπαν, θα πρέπει να διατηρήσουμε την ακεραιότητα της περιοχής του ευρώ και στη συνέχεια προσχώρησαν άλλες τρεις χώρες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άμα το δει κανείς από έξω, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αντικατοπτρίζει την τολμηρή αλλά και στεναρή ιστορική διαδικασία. Άμα δει κανείς όχι από τα μέσα το εγχείρημα αυτό, αλλά από τα έξω αυτό το οποίο βλέπει είναι δημοκρατίες οι οποίες είχαν επιλογή να παραμείνουν ή να μην παραμείνουν, αλλά και οι χώρες οι οποίες ήταν υποποίηση και αυτές που δεν ήταν υποποίηση, όλες από κοινό αποφάσισαν να διατηρήσουν τη ζώνη του ευρώ και είναι πολύ σημαντικό και το θέμα της κεντρικής τράπεζας. κεντρική τράπεζα για λόγους νομισματικής πολιτικής έπρεπε να εξασφαλίσει την μετάδοση της νομισματικής τη πολιτικής. Γι' αυτό όταν ήμουν εγώ πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, <clears throat> επενέβημε το Μάιο του 2010 στη δευτερογενή αγορά κρατικών ομολόγων, όταν δύο σχετικά μικρές χώρες είχαν προβλήματα, η Ιλλανδία, η Ελλάδα, αλλά και η Πορτογαλία. Και όταν ήμουν πρόεδρος τον Αύγουστο του 2011 και πάλι παρενέβησαν για, παρενέβημεν για δύο σημαντικές χώρες, στην Ιταλία και την Ισπανία, με ερεσιμότητα πάντα και για λόγους νομισματικής πολιτικής. Αλλά αυτό είναι ο τελευταίος λόγος που θέλω να σας αναφέρω. Χωρίς τους τρεις πρώτους λόγους δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Χρειάζεται όμως και ένα τέταρτο λόγο, αυτό που ανέφερα, για να εξηγήσετε γιατί υπήρξε αυτή η κρίση η οποία είναι πολύ πιο θετική τώρα. Τούτου λεχθέν αυτός. Όπως σας είπα προηγουμένως, δεν πρέπει να χαλαρώσουμε τις προσπάθειές μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως περιοχή του ευρώ, γιατί πρέπει να εφαρμόσουμε με αυστηρότητα τη νέα μορφή διακυβέρνησης για τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιτύχουμε την εδραίωση της ε, ενίας αγοράς και τις διαφορετικές αλλαγές δώσουμε το λόγο πάλι στο κρατήριο. μα, μια που με Ιρλανδία αναφέρατε τη χώρα μου, γιατί καμιά φορά ε, δίνω μια ρόδινη εικόνα ότι δηλαδή αναδύθηκε η Ιρλανδία, βγήκε από τη λιτότητα, ξέφυγε την Τρόικα, αλλά όμω, κύριε Τρισέ, ε, συνεχίζουν οι τράπεζε και είναι βυθισμένε στο χρέο, ε, κρατικό, δημόσιο το χρέο. Και ε, ο κόσμο θα πει ότι εσείς παίξατε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τότε που έγιναν σχετικέ συμφωνίες για την Ιρλανδία. Θεωρείτε ότι ιδίω οι μικρές χώρες ε, σαν την Ιρλανδία ε, προσπαθούν να προοδεύσουν οικονομικά και άρα μήπως κάτι θα πρέπει να γίνει με αυτή την κληρονομιά του χρέου. Κάτι θα πρέπει να γίνει, ε, αν όχι να αναδιαγραφεί το χρέο, αλλά μήπω θα πρέπει να, να παραταθεί η αποπληρωμή του γιατί τα επιτόκια είναι ε, τραγικά. Κοιτάξτε να δείτε, λέει ο Τρισέ, μετά την κρίση της Lehman Brothers Στου αμέσω επόμενου μήνες και χρόνια που ακολούθησαν από τη Lehman Brothers όλες οι χώρε αποφάσισαν και ήταν η πρώτη δηλαδή που το αποφάσισε να ε, να πούν ότι δεν θα εγκαταλείψουν τις τράπεζες. Τώρα βρισκόμαστε σε τελείως διαφορετική φάση, σε ένα άλλο σήμα, σε άλλο πλανήτη. Τώρα είναι πιο στέρεο το σύστημα. Και αυτό το οποίο θέλουμε είναι να το θωρακίσουμε τόσο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποια διάσωση. και η Ιρλανδία και οι άλλες χώρες τότε αποφάσισαν ότι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τις τράπεζες, να πέσουν έξω. Και αυτό ίσχυε και για τη Γερμανία και για την Ιταλία και για τη Γαλλία και για το Βέλγιο, για τις κάτω χώρες και για την Ιρλανδία επομένω. Αυτό είναι κάτι το οποίο κανείς θα πρέπει να το χωνέψει. τότε που ήταν επικείμενο ο κίνδυνο του να πέσει έξω το όλο σύστημα και σε εθνικό και σε διεθνέ επίπεδο, ε, τότε θα έπρεπε να ληφθούν τέτοιε αποφάσει. Αν θέλετε να σα το εξηγήσω περαιτέρω, σε άλλη στιγμή. Ναι, αλλά τέλο πάντων τι γίνεται με αυτό το χρέο τώρα που κληροδοτήθηκε. Γιατί τώρα, και τότε λίγο προ τα πίσω, θα πρέπει να δούμε το ότι. Ε, τι, το τι τοποθέτηση έχετε εσεί για για αυτό το χρέο. Εννοείται το κρατικό, λέει ο κ. Ναι, ναι, βεβαίω. Ε, καλά, ε, εννοείται ότι εάν το κράτο αρνείται, αποκρούει την οφειλή του, τότε δεν μπορεί να δανειστεί ούτε δεκάρα. Ε, αυτό είναι αυτονόητο. Γιατί όλα είναι θέμα εμπιστοσύνη. Και τώρα γινόμαστε μάρτυρε του εξή. Το ότι οι παγκόσμιοι αποταμιευτέ και επενδυτέ ξαναδείχνουν εμπιστοσύνη. Στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία και σε μερικές περιπτώσεις και προς την Ελλάδα δείχνουν εμπιστοσύνη. Και αυτό είναι το πιο πολύτιμο. Θα πρέπει επομένω να γίνει ό,τι είναι δυνατόν τόσο ώστε να ενισχυθεί αυτή η εμπιστοσύνη και να αυξηθεί αυτή η εμπιστοσύνη και αυτό θα αντικατοπτρίζεται και στα spreads. Κύριε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Για ένα άλλο θέμα, αν μου επιτρέπετε. Δεν νομίζετε ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν κάποιες κυρώσεις αυστηρότερες προς την Ρωσία. Πόσο ισχυρή είναι η Ευρώπη σε επίπεδο οικονομίας. Ποιες, ποια είναι τα δύνατα, τα τρωτά μας σημεία. of... Uh, Τρισέ, ε, νομίζω ότι αυτό δεν είναι δικό μου θέμα να σας το απαντήσω είναι το τρέχουσες οι εξελίξεις αυτές, αλλά μπορώ απλώς να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου όλα αυτά καταδεικνύουν ότι όλοι όσοι ισχυριζόντουσαν πως η σταθερότητα και η ειρήνη, όχι μόνο στα οικονομικά, γενικότερα, ότι επομένως αυτά ήταν δεδομένα αγαθά Τώρα πρέπει να αναθεωρήσουν. Γιατί, κοίταξτε, δεν ε, τα σκέφτομαι απεσιόδοξα. Απλώς, τι να σας πω. Ξέρετε, ε, η γυναίκα μου είναι ουκρανικής καταγωγής. Και τα παιδιά μου επομένως είναι μισή Ουκρανή. Άρα με καίει το τι γίνεται στη χώρα. Πάντως, σας λέω και πάλι. από περιέργεια έξα μια ματιά σε μια πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρετε ότι κάθε έξι μήνες γίνεται μια εμπεριστατωμένη έρευνα και πάντοτε τα ερωτήματα είναι τα ίδια. Σε αυτό το ερωματολόγιο λοιπόν είπαν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα εξή. Και σας λέω επιλέξει ποια ήταν η φράση που θα πρέπει να πει συμφωνώ ή διαφωνώ. Θα μπορούσε μια κοινή άμυνα και κοινή ασφάλεια στην Ευρώπη. Γιατί για την ε, Ευρωζώνη ε, θα μπορούσε να υπάρχει και 73% συμφώνησε και 19% διεφώνησε επομένω αυτή η αίσθηση του ότι βρισκόμαστε σε έναν κόσμο, οπότε θα πρέπει να έχουμε μια αίσθηση ταυτότητας και ότι θα πρέπει να έχουμε μια κοινή ασφάλεια και άμυνα, αυτό ισχύει και με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Και αν έχει κανείς μια ματιά ε, στο τι απαντήθηκε αναχώρα, θα δείτε ότι η απάντηση ήταν η ομοιογενής σε όλες τις χώρες. Και αυτά πριν τα γεγονότα στην Ουκρανία. Τέλη του 2013 έγινε αυτή η έρευνα, αυτό το γκάλωπ συμφωνία και διαφωνία όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση με ενιαίο νόμισμα το ευρώ. Εδώ έχουμε μια ελαφρά πλειοψηφία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στην Ευρωζώνη είναι συντριπτική η πλειοψηφία υπέρ του ευρώ. 71% συμφώνησε με το ευρώ στη Γερμανία. Διαφωνεί το 25%. Στη Γαλλία 63% συμφωνούν και 32% διαφωνούν. Να, ε, τώρα απαντώ και τις προηγούμενες ε, ερωτήσεις. Και μετά για να επαληθευθεί η απάντηση, για να δούμε ε, εάν κατανόησαν την ερώτηση. Οι Βρετανοί τι είπαν, 19% όχι, 14% ότι διαφωνούν. 19% θέλουν το ευρώ, 74% όχι. Ήταν αυτή η εμπειρία του. Αλλά όμω στην Ευρωζώνη συμφωνούσαν όλοι. όλοι. Κατά πλειοψηφία. Βλέπετε. Κάθε θα κανείς ε, την στάση τη μειοψηφία να την ε, ε, σχολιάσει, να την εξηγήσει, αλλά πάντω έχουμε ουσιαστικά δύο τρίτα που συμφωνούν με το ευρώ στη Γερμανία και στην δική μου χώρα. Αυτό σημαίνει ότι κατάλαβαν την ερώτηση. Εσείς κύριε. Team από την Γερμανία. Στην Wirtschaftswoche εργάζομαι οικονομική εφημερίδα. Θέλω να μου πείτε τι άποψη έχετε για ένα πιθανό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακούγεται πως μπορεί να αρχίσει να αγοράζει ομόλογα όχι μόνο κρατών της Ευρωζώνης αλλά ίσως και εταιριών και ίσως και ομόλογα είπα. Θεωρείτε πως ε, είναι μια καλή ιδέα να εξασθενήσουμε το νόμισμά μας και να αντισταθούμε στον αποπληθωρισμό που υπάρχει στον Νότο και ποιες είναι οι τυχόν αρνητικές πτυχές του προγράμματος. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα σέβομαι πλήρως τους ε, συναδέλφους μου του ΔΣ της ε, τράπεζας και δεν θέλω να παρέμβω στις αποφάσεις τους. Πρώτη παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη πρέπει να αντιληφθούμε και το εξηγώ αυτό παντού γιατί δεν είναι εύκολο να είναι αντιληπτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρει μια ασφάλεια σε όλες τις ε, τράπεζες της Ευρωζώνης ότι θα έχουν όλη την απαιτούμενη ρευστότητα σε περίπτωση ανάγκης με σταθερό επιτόκιο, κάτι το οποίο εισήχθη για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2007 όπως ανέφερα, 95 δισεκατομμύρια που δόθηκαν τότε και γενικεύθηκε μετά την Lehman Brothers και εξακολουθεί να υπάρχει. Οπότε οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα στην Ευρώπη έχει πρόσβαση σε όλη τη ρευστότητα που χρειάζεται, αρκεί βεβαίω να δώσει κάποιες εγγύησεις. Ε, αυτό σημαίνει πως μπορούν να λάβουν 3-4 φορές την ε, ρευστότητα την οποία ζητάνε αυτή τη στιγμή σε περίπτωση ανάγκης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αντιληφθούμε γιατί είναι λίγο πολύ το ισοδύναμο αυτού που κάνουν οι ΙΠΑ. Οι ΙΠΑ έχουν μια οικονομία η οποία βασίζεται στις αγορές για τη χρηματοδότησή της, 80% αγορές, 20% τράπεζες. Οπότε η κεντρική τράπεζα εκεί τροφοδοτεί τις αγορές ε, με την αγορά δημοσίων και ιδιωτικών αξιογράφων γιατί είναι το βασικό κομμάτι της ε, χρηματοδότησης της οικονομίας στην Ευρώπη. Οι τράπεζες χρηματοδοτούν κατά 80% την οικονομία και 20% οι αγορές και βεβαίως δεν προξενεί εντύπωση το ότι η ρευστότητα πάντα επικεντρωνόταν στις τράπεζες με, όπως είπα ξανά, αυτή την εξασφάλιση που δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μπορούν να έχουν όση ρευστότητα χρειάζεται. Βεβαίως αυτό δεν μας εμπόδισε να αγοράσουμε εμείς αξιόγραφα, όπως ξέρετε. Αυτό το κάναμε και για δημόσια αξιόγραφα τον Μάιο του 10 και Αύγουστο του 11 και συναλλαγές αυτές, όπως είπαμε, είναι αν θέλετε ένα είδος εξασφάλισης, εάν χρειαστεί και εάν ζητηθεί και βέβαια και τα ίδια τα κράτη συμμετέχουν και πρέπει να σας πω πως ε, εγώ το διαπραγματεύτηκα αυτό με τους επικεφαλής των κυβερνήσεων τον Ιούλιο του 2011, αλλά το του Λεχθέντος επίσης είχαμε αγοράσει και στο παρελθόν και ιδιωτικά ε, αξιο αξιόγραφα. Ε, υπήρχε δυνατότητα, το κάναμε. Θα δούμε λοιπόν τι θα συμβεί. Εγώ θεωρώ πως ε, δεν αποκλείεται, αλλά και πάλι ε, δεν έχω κάποια συμβολή να δώσω τώρα στην Κεντρική Τράπεζα, αλλά δεν αποκλείεται ειδικά να υπάρξει αγορά ιδιωτικών αξιογράφων για να βοηθήσουμε να να ζωογονηθούν οι αγορές οι οποίες δεν λειτουργούν καλά αυτή τη στιγμή και μιλάω ιδιαίτερα για την τιτλοποίηση, για την τιτλοποιημένη αγορά η οποία είχε πεθάνει μετά την κρίση και μπορεί να χρειαστεί να επανέλθει στη ζωή για να ανακουφιστούν λίγο οι τράπεζες από το βάρος και να χρηματοδοτηθούν ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάτι άλλο το οποίο επίσης δεν αποκλείεται θα ήταν να διακοπεί σταδιακά ή εντελώς η αδρανοποίηση του προηγούμενου προγράμματος ε, σταθερότητας που είχε γίνει επί εποχής μου και να μην υπάρχει αυτή η ουδετερότητα η οποία θα υπήρχε και σταδιακά να αποσυρθεί αυτή η ρευστότητα. Βεβαίω το βασικό πρόβλημα είναι πως πρέπει να είμαστε σίγουροι γιατί λέτε πως ε, ε, είχαμε θέσει ως στόχο το να αποφύγουμε τον πληθωρισμό μα να αποφύγουμε και τον πληθωρισμό και τον αποπληθωρισμό είχαμε ως στόχο αυτό το οποίο λέμε εμείς ε, σταθερότητα τιμών είναι λιγότερο από δύο αλλά κοντά στο δύο και μάλιστα τα 15 πρώτα χρόνια του ευρώ ήμασταν στον ετήσιο πληθωρισμό γύρω στο 2% ευθυγραμμισμένη με τον ορισμό της σταθερότητας τιμών. Και σας έχω μία αποκάλυψη εδώ. Ο ορισμός της σταθερότητας των τιμών αυτή την στιγμή είναι πρακτικά ο ίδιος στην Ιαπωνία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ και στην Ευρωζώνη. 2% παντού, ε, μέσω μακροπρόθεσμα. Και όπως σας είπα για εμάς είναι κάτω αλλά κοντά στο 2 κάτω από το 2 αλλά κοντά στο 2 και η... τα νομίσματα που είναι στο καλάθι των ειδικών τραβηθικών δικαιωμάτων του Δουνουτού έχουν όλα τον ίδιο ορισμό της σταθερότητας τιμών που σημαίνει όχι πληθωρισμός ε, μεσομακροπρόθεσμα, όχι πληθωρισμός Κοντά στο 2 και 2. Αυτό ε, είναι από πέρσι, είναι νέα εξέλιξη. Αυτή η σύγκληση δηλαδή ε, είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό για εμένα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τρισέ μπορεί να μείνει για 15 λεπτά. Ε, αν ε, θέλετε να θέσετε ερωτήματα, ξεκινάμε τον γύρο και μετά έρχομαι από την άλλη πλευρά της αίθουσας για όσους έχουν ερωτήματα. Παουλούχα από την Πορτογαλία. Ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα. Τι σχόλια έχετε για την καθαρή έξοδο της Πορτογαλίας από την διαδικασία σταθεροποίησης. Πώς θα περιγράφατε λοιπόν την έξοδο της Πορτογαλίας. Με έχουν ερωτήσει πολλές φορές αυτό το ίδιο ερώτημα. Για μένα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση η οποία ελήφθη και έχω πει πάντα ότι κατά τη μου άποψη ήταν μια κρίση που εναπέκειτο στην πορτογαλική κυβέρνηση επί τη βάση όλων των πληροφοριών που είχε η πορτογαλική κυβέρνηση, ιδίως σε ό,τι αφορούσε το επίπεδο εμπιστοσύνης που είχε επιτευχθεί μετά από την προσαρμογή, η οποία ήταν δύσκολη, πρέπει να το πω, πολύ δύσκολη, αλλά απόλυτα απαραίτητη και ήταν επιτυχής. Όταν δω λοιπόν τι έγινε στην Πορτογαλία και πώς την έκρινε ο υπόλοιπος κόσμος, ήταν μια επιτυχής προσαρμογή. Αυτή λοιπόν ήταν μια απόφαση της πορτογαλικής κυβέρνησης, την οποία σέβομαι απόλυτα. Ευχαριστώ. Ο κύριος πίσω, ναι, από τη Σλοβενία. Ο πληθυσμό τώρα είναι πολύ χαμηλότερος από τον στόχο του 2%. Μήπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να λάβει υπόψη προβλήματα όπως η ανεργία και η έλλειψη οικονομικής ανάπτυξης και όχι μόνο τον πληθωρισμό. Και η πολιτική λιτότητας πιστεύω ότι είναι κάτι το λανθασμένο. Δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο από θεσμούς όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τώρα που δεν χρειάζεται να σας τόσο προσεκτικός με τα λόγια σας, ποια είναι η κρίση σας για τις πολιτικές αυτές που ακολουθήθηκαν. Όπως είπα, πρώτα απ' όλα λέει ο κύριος Τρίσε, δεν θέλω να σχολιάσω τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν σε χώρες που είχαν προβλήματα και δεν θα τις ονόμαζα πολιτικές ε, λιτότητος. Ήταν μια επανόρθωση των ανισομεριών, των ανισορροπιών. Εάν δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα είχε υπάρξει, αν δεν είχε, είχαν δημιουργηθεί αυτές οι ανισομέρειες, δεν θα υπήρχε ανάγκη για πολιτική λιτότητα και εξάλλου. Δεν ήταν πολιτική λιτότητα. Όταν κανείς έχει μεγάλες ανισομέρειες και ζητάει από τον υπόλοιπο κόσμο να σε χρηματοδοτήσει και δεν μπορεί να σε χρηματοδοτήσει ο υπόλοιπο κόσμος ή δεν θα έχει κανείς καμιά βοήθεια σε αυτό ή θα έχει κάποια βοήθεια. Κάποια βοήθεια όμως σήμαινε ότι θα έπρεπε οι χώρες αυτές να εξασφαλίσουν την αξιοπιστία τους στο δρόμο προς την ανάκαμψη. Όλες οι εμπλεκόμενες χώρες το έκαναν αυτά, όπως όλος ο κόσμος το, το γνωρίζει. Για το άλλο ερώτημα που αναφέρεται για το χαμηλό επίπεδο του πληθωρισμού, η δική μου κατανόηση και πάλι είναι ότι περνάμε μια χρονική διάρκεια χαμηλού πληθωρισμού που είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο για πολλούς λόγους. Στην Ευρώπη έχουμε ένα πρόσθετο λόγο που είναι ότι για τις χώρες οι οποίες έχασαν την ανταγωνιστικότητά τους πρέπει να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ελέγξουν τα εισοδήματα, το κόστος των δημοσίων δαπανών, τον εθνικό προϋπολογισμό για να μπορέσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπω ως απόλυτα φυσιολογικό. Αν δούμε τη ζώνη του ευρώ σαν σύνολο, οι αρχές που είναι αρμόδιες για το σύνολο της ε, ζώνης του ευρώ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αφενός αλλά και το ευρωπαϊκό επίπεδο από την άλλη μεριά θα πρέπει να εξετάσουν αν σε χώρες οι οποίες έχουν περιθώριο ελιγμών έχουν γίνει οι σωστές ενέργειες για να εκμεταλλευτούν αυτό το περιθώριο ελιγμών που θα επέτρεπαν να έχουμε σαν μέσον όρο ε, ένα μεγαλύτερο ποσοστό πληθωρισμού στην περιοχή του ευρώ. Σίγουρα πρέπει να αποτρέψουμε την αποσταθεροποίηση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό. Γιατί όλες οι προσδοκίες στη ζώνη του ευρώ για τον πληθωρισμό ε, ε, έπαιζαν κάποιο μεγάλο ρόλο στην λειτουργία της οικονομίας. Επομένως, δεν έχει πάψει να έχει κανείς την ε, στάση αυτή ότι θέλουμε τον πληθωρισμό να είναι κοντά στα 2% και λίγο λιγότερο από τα 2% και για την ε, τωρινή κατάσταση με το χαμηλό πληθωρισμό εγώ πιστεύω ότι θα λειτουργήσει η οικονομία της αγοράς σε οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν 6-7% πλεόνασμα στο τρέχον ισοζύγιο κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει και σε περισσότερες επενδύσεις, μεγαλύτερες αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια, όπως βλέπουμε τώρα να λαμβάνει η χώρα και πιστεύω ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η οικονομία της αγοράς στις χώρες αυτές και δεν μιλάω μόνο για τη Γερμανία, αλλά για όλες τις χώρες που έχουν πλεονασματικό ισοζύγιο τρέχουσών συναλλαγών. Ελπίζω λοιπόν ότι έχω απαντήσει και στο δικό σας ερώτημα αφού απάντησα στο ερώτημα του πρακτέου σε σχέση με τις νέες αποφάσεις που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα και έχω ε, απόλυτο σεβασμό για τη σοφία του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γιάννης Ρέγμαν από την ε, Δανία. Μήπως θα μπορούσατε να κοιτάξετε λίγο πιο μπροστά και κύριε Τρισέ να μας δώσετε και κάποιες συμβουλές. Σε λίγε εβδομάδε γίνονται ευρωεκλογέ. Μία από τι προκλήσει που θα αντιμετωπίσει το νέο κοινοβούλιο και η νέα Κομισιόν είναι το θέμα τη ανεργία, ιδίω τη ανεργία των νέων. Και μα ενδιαφέρει ποια θα είναι η μελλοντική πορεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά. Πώ θα συμβουλεύατε λοιπόν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβερνήσεις για να έχουν περισσότεροι άνθρωποι στην Ευρώπη δουλειά και ιδίως νέοι. Ποιες θα είναι οι συμβουλές σας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα. Πρώτα απ' όλα, να σας πω ότι βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είσαστε, δημοσιογράφοι, δεν είσαστε βουλευτές, είσαστε δημοσιογράφοι. Αλλά ας πούμε ότι ήσασταν εκπρόσωποι των λαών της Ευρώπης, ότι ήσασταν βουλευτές ότι είχατε αυτή την νομιμοποίηση λόγω της άμεσης καθολικής εκλογής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη δική μου άποψη στο μέλλον, θα πρέπει να διαδραματίσει ένα πιο σημαντικό ρόλο. Γιατί είναι μεταξύ των θεσμικών αυτών οργάνων το θεσμικό όργανο που είναι δημοκρατικά ε, υπόλογο. Στο Κίελο, στη Γερμανία, είχα κάνει μια σειρά προτάσεις σε μια ομιλία για την δυνητικότητα να υπάρξει μια οικονομική και δημοσιονομική ομοσπονδία σε εξαιρετικό επίπεδο. Η ιδέα είναι πολύ απλή. Αν εφαρμόσετε τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και γίνονται αυτές οι συστάσεις σε μια χώρα που δεν τις εφαρμόζει και πάλι μια δεύτερη φορά δεν τις ε, ε, εφαρμόζει και υπάρχει διαφορά απόψε μεταξύ της θέσης της Κομισιόν και του Συμβουλίου και της χώρας αυτής. Θα πρέπει να μπορεί να πει μια χώρα ότι εγώ είμαι σε αντί, αντίρρηση α, με τις συστάσεις αυτές και ζητώ την τελική θέση του Κοινοβουλίου. Φυσικά θα πρέπει να είναι το Κοινοβούλιο που να περιλαμβάνει μονάχα τους βουλευτές που είναι μέλη της ζώνης του ευρώ. Γιατί όλοι πράγματι εμπλέκονται και αν δεν υπάρξει σωστή λειτουργία μιας χώρας αυτό δημιουργεί πρόβλημα για το σύνολο του συστήματος. Δεν θα ήταν λοιπόν παράλογο να ζητήσουμε την τελική απόφαση να ληφθεί μαζί με τα Εθνικά Κοινοβούλια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι μια ιδέα λοιπόν που εγώ διατύπωσα και νομίζω ότι λαμβάνει υπόψη και την αρχή της επικορικότητας γιατί θα λειτουργούσε μονάχα σε έκτακτες περιστάσεις με την αρχή της αποτελεσματικότητας και σε τελική ανάλυση με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να γίνει αυτή η απόφαση από τους δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους των λαών. Και τώρα για τους νέους που λέτε, για την ανεργία των νέων. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ στο να δημιουργήσουμε μία ε, νέα ισορροπία, αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε δημιουργία απασχόλησης με πιστικό τρόπο. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και για μένα αυτό εξαρτάται από το να έχουμε μια πολύ καλή ισορροπία και να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις. Αν δείτε σε κάποια χώρα να υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της ε, απασχόλησης για τους νέους και γενικά για τον πληθυσμό, τότε αυτό σημαίνει ότι έχετε μεγάλες ανισομέρειες στο επίπεδο της αγοράς εργασίας. Αν έχετε καλή δομή στην αγορά εργασίας, τότε θα έχετε την ίδια ανεργία και για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Μπορεί να μην είναι χαμηλή, γιατί όλοι είχαμε προβλήματα ανεργίας, αλλά θα είναι ενιαία μορφής η ανεργία. Είναι απαραίτητο Ξεχάσαμε το πρόγραμμα 2020 ε, στη τη της τη Λισαβόνα θα πρέπει να υλοποιηθεί, γιατί αυτό είναι ο πιο αποτελεσμό τρόπο ούτω ώστε να εκμεταλλευτούμε τι δυνατότητε τη Ευρώπη στο σύνολό του. Και μην ξεχνούμε, μιλούμε για τους 28 αλλά κυρίως τις δυνατότητες της Ευρωζώνης. Εκεί επιμένω διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις, τήρηση της νέας αποτελεσματικής διακυβέρνησης και δημοκρατική νοημοποίηση και ακόμα σήμερα το Κοινοβούλιο έχει τεραστία ευθύνη. Και αυτό θα πρέπει να το χωνέψουν οι Ευρωπαίοι. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον η επικοινωνία αποδίδει ε, όσο θα έπρεπε. Τέλος πάντων, ε, να που έχω τώρα την ευκαιρία να επικοινωνήσω με εσά που ασχολείστε με την επικοινωνία τώρα. Έχουμε το, το, ε, το, επόμενο πάνελ, αλλά πριν ε, έχουμε και άλλους που έχουν στο λόγο, ο κύριος εκεί δεξιά και εσείς εδώ μπροστά, εσείς κυρία στο μέσο μόνο της αιθούσης, ωραία, τότε να υποβάλλετε όλοι μαζί τις ερωτήσεις σας και απαντήσει όλοι μαζί σας, πειράζει κύριε Τρίσσερ, ναι, ναι, εντάξει. Ωραία, επόμενες εσείς από τη δεξιά, από τη πτέρυγα, παρακαλώ συντόμως. Ντάριο Τσιντσόνη ονομάζομαι, καλησπέρα σας από το τέταρτο κανάλι του Sky. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κατά τη γνώμη σας, στο μέλλον, φώνετε ακουστικά, σας λέω τελικά για να είμαστε επικοινωνούμε, είναι δυνατόν να ανέβει το, το 3% αυτό το κατόφλιο σε σχέση με το ε, έλλειμμα και επίσης τι γίνεται όσον αφορά ε, το, το ότι μπορεί οι ευρωσκεπτικιστές να τα πάνε καλά στις ε, εκλογές. Εδώ η κυρία στο μέσο της έδωσης. Πρώτα εσείς. Μποζονίν ονομάζομαι, προέρχομαι από την Ελλάδα και επιμένετε στο θέμα της δημοκρατικής νοημοποίησης, η ε, δε Τρόικα. Είχε κατηγορηθεί ότι ακριβώς δεν ε, είναι υπόλογη σε κανέναν και ότι ε, ε, έπραξε λάθη στην Ελλάδα. Αυτό πώς μπορεί να διορθωθεί κατά τη γνώμη σας. Και τώρα η κυρία πίσω από σας. Στη συνέχεια, προηγούμενη ερώτηση, θέλω να πω κάτι σε σχέση με την κρίση στην Ουκρανία. Τι λέτε, εάν επιδεινωθούν οι σχέσεις με την Ρωσία, αυτό θα μπορούσε να φέρει ύφεση στην Ευρώπη λόγω των εξελίξεων της, των τιμών του φυσικού αερίου. Τώρα, εσείς στην αριστερή πτέρυγα να σα ρωτήσω κάτι για τη Λατωνία στην οποία μίλησατε, από εκεί προέρχομαι, επί τη βάση τη εμπειρία σας. Ε, τα πάει καλά, τα πήγε καλά η Λετωνία όσον αφορά την προσχώρηση στην Ευρωζώνη. Τρισέ. Ε. Ναι. Σημείωσα όλες τις ερωτήσεις. Ε, για την πρώτη ερώτηση από την Ιταλία. Εάν θα αλλάξουμε το 3% αυτό ήταν το ερώτημα. Ναι, στο μέλλον. Ό, η απάντηση είναι πολύ απλή. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Νομίζω πως ε, η εμπειρία που είχαμε ήταν πάρα πολύ κακή. Δεν υπάρχει συνένεση για κάτι τέτοιο στην Ευρώπη κατά την άποψή μου για να αλλάξει το κατόφλι, το οποίο θετικά εισήγαγα εγώ στις διαπραγματεύσεις στη συνθήκη του Μαστρίχτ γιατί φαινόταν πως είναι ένα κατόφλι το οποίο ήταν απλό και το καταλάβαιναν όλοι και να σας πω πως έγινε λίγο πολύ αν θέλετε ένα παγκόσμιο μέτρο αναφοράς δηλαδή το 3% το οποίο δεν θα ξεπερνιέται παρά μόνο σε εξαιρετικές ε, περιπτώσεις. Οι διατάξεις αυτές του Συμφώνου Σταθερότητας ε, έχουν γενικευθεί θα έλεγα, αλλά δεν νομίζω πως υπάρχει συνένεση για κάτι τέτοιο. Ε, ε ξεχνάμε κάτι άλλο. Όταν ξεκινήσαμε να μην σεβόμαστε το σύμφωνο σταθερότητας για ανάπτυξη, κάτι το οποίο ξεκίνησαν οι μεγάλες χώρες ε, έναντι των μικρών και όπως σας είπα εγώ συμμετείχα στη συζήτηση από το Δεκέμβριο του 2003 ήδη, τότε υπήρχε, αν θέλετε, μία ήπια αδιαφορία για τα ζητήματα αυτά των προϋπολογισμών και οι οικονομολόγοι παγκοσμίω λέγανε πως έβαλαν ζουρλομανδία από μόνοι τους οι Ευρωπαίοι και δεν έπρεπε να περιοριστούν τόσο. Βεβαίως βλέπουμε το 2009, 10, 11, 12, 13 τι σήμαινε το ότι δεν σεβόμασταν τους εν λόγω περιορισμούς και αν δείτε τις ε, χώρες ε, που σεβάστηκαν και δεν σεβάστηκαν το σύμφωνο βλέπετε πώς ανταμείφθηκαν αυτές οι οποίες διαχειρίζονταν ε, σωστά τα δημόσια οικονομικά τους. Για τους ε, βροσκεπτικιστές θα έλεγα μόνο πως ε, ζούμε σε πολύ ζωντανές ε, δημοκρατίες, υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και εγώ πιστεύω στην Ευρώπη. Πιστεύω στο ιστορικό αυτό οικοδόμημα και νομίζω πως υπάρχει μια συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που εμπιστεύονται την Ευρώπη και σε πολλές ε, διαστάσεις ε, θα αναφέρω και αυτήν στην οποία υπάρχει λιγότερη πρόοδος την ασφάλεια και την άμυνα και όμως ε, υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία υπέρ οπότε εγώ αναμένω να εξηγήσουν αυτοί οι άνθρωποι την ε, θέση τους ε, στους ε, πολίτες της Ευρώπης. Αυτή είναι η απάντησή μου. Για την Τρόικα και την Ελλάδα. Να σας υπενθυμίσω, να μας υπενθυμίσω. Πώς η Τρόικα αποτελείται από ποιους. Τον εκπρόσωπο του Δούνου του. Οι χώρες στην Ευρώπη ζήτησαν από την διεθνή κοινότητα να τις βοηθήσει η διεθνής κοινότητα, δηλαδή η Ινδία, η Κίνα, η Βραζιλία, Μεξικό και η Λιπή, συν όλες οι ανεπτυγμένες οικονομίες, η Ιαπωνία, ΗΠΑ και Ευρώπη. Πρέπει να πιστούν πως δανείζουν χρήματα σε μια χώρα η οποία θα τα εξοφλήσει και θα είναι φερέγγια, αλλιώ δεν έχει νόημα. Οπότε ε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Το ίδιο και η Κομισιόν. Η Κομισιόν πρέπει να πείσει όλα τα κοινοβούλια της Ευρώπης. Τα, κοινοβούλια που εκπροσωπούν τους λαούς της Ευρώπης. Οπότε στις διάφορες πρωτεύουσε κρίνουν το εάν είναι σωστό ή όχι να δανείσουν λεφτά. Οπότε μπορεί να παρουσιάζεται την Τρόικα ως σκληρή και υπερβολικά δύσκολη στις συζητήσεις, αλλά και πάλι. Αν δεν θέλετε δύσκολες συζητήσεις, ε, μπορείτε πάντα να μην ε, ζητήσετε βοήθεια. Είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία πρέπει να αντιληφθούμε λίγο ποια είναι η θέση μας. Ε, εμείς ήμασταν παρατηρητές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι παρατηρητής, δεν αποφασίζει ούτε στις Βρυξέλλες ούτε στην Ουάσιγκτον. Και βλέπαμε τις δυσκολίες ε, μία τέτοιας κατάστασης προσαρμογής που είναι πάντα εξαιρετικά δύσκολη. Οπότε το μάθημα είναι να μην βρεθείτε σε ε, κατάσταση με έλλειμμα 15%. Ε, τότε ελήφθησαν οι φρικτές αποφάσεις. Όχι όταν φτάνει η ώρα να διορθωθούν επειδή πρέπει. Και βεβαίως η χώρα έχει πάντα την δυνατότητα να δει από μόνη της την προσαρμογή και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προστατεύσει τις θέσεις εργασίας στην προσαρμογή. Ε, εκεί πέρα νομίζω πρέπει οι πανεπιστημιακοί οικονομολόγοι να το δουν περισσότερο. Εάν, ελπίζω να μην γίνει, στο μέλλον κάποιες χώρες ε, πρέπει να επανέλθουν στην ομαλότητα από μια πάρα πολύ ανώμαλη κατάσταση οι οικονομολόγοι της χώρας βεβαίως αλλά και στο επίπεδο θα έλεγα του, της ακαδημαϊκής συνένεσης πρέπει να δουν πώς θα προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας και όχι μόνο το εισόδημα όσων έχουν δουλειά έτσι, γιατί βεβαίως αυτοί θέλουν να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους και έχουν περισσότερη διαπραγματευτική ισχύ από τους νέους που χτυπάνε να μπουν στην αγορά εργασίας. Έτσι. Ναι, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από κοινωνική σκοπιά. Τώρα για την Ουκρανία δεν θα επεκταθώ. Δεν ναι, προσθέσω τίποτα. Σε αυτά τα οποία είπα είναι μια κατάσταση για την οποία ελπίζω επειδή ζούμε σε καιρούς επικίνδυνους και δύσκολους ελπίζω η διεθνής κοινότητα να βρει έναν τρόπο να διατηρήσει την ε, ανεξαρτησία της χώρας, την οποία γνωρίζω, και βεβαίω την ειρήνη και τη σταθερότητα στο μέρος αυτό της Ευρώπης. Ε, αυτό δεν ισχύει ε, τα ευρωπαϊκά μου πιστεύω. Όσον αφορά την Λετωνία, η Λετωνία είχε συνδεθεί πολύ στενά με το ευρώ το, το νόμισμά της ε, και είχε βεβαίως δραματικά προβλήματα όπως όλες οι βαλτικές χώρες αλλά κατάφερε να διατηρήσει την δημοσιονομική σταθερότητα σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες χωρίς να ζητήσει βοήθεια κάτι το αξιοθαύμαστο και πραγματικά νομίζω πως αυτό είναι ε, επιτυχής ε, προσαρμογή, πάντα δύσκολη γιατί όπως είπαμε η φοιτηρία ήταν πάρα πολύ δύσκολη αλλά θα έλεγα πως ο τρόπος με τον οποίο οι βαλτικές χώρες βρήκαν τρόπους μέσα στην κρίση να μην φτάσουν σε φρικτές αναταραχές ε, νομίζω ήταν ε, αξιοθαύμαστος. Σας ευχαριστούμε κύριε Τρισέ. Νομίζω πως Θέλατε να μιλήσετε σύντομα για την έκθεση της Τριμερούς Επιτροπής που δημοσιεύτηκε σήμερα ή στο Ευρωπαίος Πρόεδρος και ειδικά για μια πρότασή της που αφορά την διασφάλιση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πρέπει να γίνει πιο σημαντικός. Πράγματι. Είναι σύμπτωση ε, η Τριμερής Επιτροπή στο επίπεδο Ευρώπης και σε παγκόσμιο επίπεδο είχε εξετάσει τα της Ευρώπης δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας επί Μάριο Μόντι όταν ήταν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πυλώνα της τριμέρους αυτής ομάδας και ξεκίνησε τις εργασίες της όταν η κρίση ήταν δραματική και σήμερα δημοσιεύουμε την έκθεση που είναι νομίζω ενδιαφέρουσα. Γιατί υπάρχει αν θέλετε σκοπιά πολλών ανθρώπων όπως ε, Σκοαό, ε, πρώην Πρωθυπουργός Φιλανδία, ο Αλφοντερίε, Υπουργό Οικονομικών τη Γαλλίας, ο Ότμαρ Ισινγκ, ε, φίλος μου, ο Τζον από την ε, Βουλή των Λόρδων, Αντρέης Ολεσόφσκι, πρώην Υπουργό ε, Εξωτερικών και Οικονομικών ε, της Πολωνίας, Φερνάντο ο Χάνς Φίγερς από την ΣΕΛ, ο Αντρέ Σαπίρ, πολύ γνωστός στις Βρυξέλλες, εισηγητής ήταν και ο Πόλεβεο. Ευρωπαίος Διευθυντής. Έχουμε λοιπόν μία ανάλυση της κατάστασης, ε, ε, εκτιμούμε τα όσα έγιναν ε, και ζητάμε να αναπτυχθεί αν θέλετε μία ευρωπαϊκή διήγηση σε πέντε άξονες. Ο σεβασμός της αρχής επικουρικότητας, η οικονομική και δημοσιονομική διακυβέρνηση με στόχο της δημιουργία θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της μαζικής ανεργίας που γνωρίζετε πως υπάρχει σε πολλές χώρες, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, το ανέφερα ήδη, ε, σύμφωνα με τα όσα λέει η ατζέντα της Λισαβόνας και το 2020. Επίσης, αναφέρουμε με αρκετά μεγάλη συνένεση την ε, σταθεροποίηση, ειρήνη, ασφάλεια εσωτερική και εξωτερική. Ε, νομίζω το ζητάνε αυτό οι Ευρωπαίοι. Και τέλος ε, ο, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πρέπει να γίνει πιο σημαντικός από ποτέ πέραν από τον έλεγχο του προϋπολογισμού είναι το μόνο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που έχει δημοκρατική νομοποίηση που προέρχεται από την άμεση καθολική ψηφοφορία ε, η οποία βεβαίω ε, ε, τονίζεται και θα παίξουν εδώ πέρα κέριο ρόλο οι ευρωεκλογές του 2014. Αυτά είναι τα βασικά. αν θέλετε γραπτό και όχι ηλεκτρονικό το έγγραφο έχω και κάποια αντίγραφα τα αφήνω εδώ ελπίζω λοιπόν όπως ε, είπα να μην σας έφαγα πολύ χρόνο ήταν μεγάλη μου χαρά που ήμουν εδώ σήμερα και είμαι στη διάθεσή σας για συζητήσεις αν θέλετε διμερείς σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε Σας ευχαριστούμε, ήσασταν καταπληκτικός, μοιραστήκατε μαζί μας τις θέσεις σας και τον χρόνο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Um, Μια σύντομη διακοπή για 15 περίπου λεπτά και θα ξαναβρεθούμε για τη συζήτηση μεταξύ των βουλευτών.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

Okay, Κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη φάση της ε, συνεδρίασής μας το απόγευμα. Παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας, καθίστε στις θέσεις σας, θα ξεκινήσουμε και θα, έρθουνε, θα έρθει και ένας ακόμα βουλευτής ε, σε λίγο. Καθίστε λοιπόν παρακαλώ. Okay, so... Εντάξει. Αν μπορώ να έχω την προσοχή σας λοιπόν, γιατί αλλιώς θα είναι πολύ δύσκολα, αν μιλάτε και κάνετε πηγαδάκια. Παρακαλώ κυρία μου, σας παρακαλώ ευχαριστώ, αν μπορώ να έχω την προσοχή σας. Εντάξει. Το τμήμα αυτό λοιπόν έχει να κάνει με τις πολιτικές ατζέντε και τις επιλογές των ψηφοφόρων για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Πολλοί από εσά έχετε ερωτήματα τα οποία θέλετε να θέσετε στο πάνελ μας. Έχουμε τέσσερις βουλευτές. Τρεις ε, δεν θα κατέβουν στις εκλογές και ένας βουλευτής θα διεκδικήσει και πάλι την έδρα του. Έχουμε τον Μάτιου Γκρός, από την ομάδα του ΕΛΚ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι Βέλγος Ευρωβουλευτής, τον Ερίκε ε, Σαλόμ από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών από την Ισπανία. Θα έρθει η Ζαμπέλ από τους Πράσινους εδώ στο Βέλγιο και έχουμε επίσης μαζί μας τον Γιούργεν Κλούτε από την ομάδα της Γκουε, την αριστερή ενωτική ομάδα στην Ευρώπη και είναι Γερμανό. Ένα μονάχα ερώτημα θέλω να δώσω σε όλου του βουλευτέ και στη συνέχεια είναι η δική σα ε, σειρά να θέσετε ερωτήματα. Να θέσετε λοιπόν ερωτήματα τα οποία μπορεί να είναι σημαντικά για εσά ω δημοσιογράφου και ω προερχόμενοι από χώρες οι οποίε δεν θα έχουν ενδεχομένω μεγάλη προσέλευση στι ευρωεκλογέ. Αν μπορώ λοιπόν με εσά κύριε Γκρός να ξεκινήσω Υπάρχει το σύνθημα για τις ευρωεκλογέ. Αυτή τη φορά είναι διαφορετικά αυτό είναι το σύνθημα. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τώρα πολύ μεγαλύτερη σημασία για τους ψηφοφόρους λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας. Έχουν περισσότερες εξουσίες οι ευρωβουλευτές. Πιστεύετε ότι αυτό το μήνυμα είναι κάτι το ακουστό από τους πολίτες μας. Μπορώ να μιλήσω ό,τι γλώσσα θέλω. θα μιλήσω γερμανικά λοιπόν ως καλός Βέλγος. Λοιπόν, κοιτάξτε, είμαι Βέλγος, ε, γερμανόφωνος από τα σύνορα εκεί με την Γερμανία και το αυτό το οποίο βλέπω εγώ τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη είναι πως ειδικά στις μεθοριακές περιοχές ε, είναι πως ο κόσμος έχει πολύ περισσότερες και υψηλότερες προσδοκίες από αυτά τα οποία κάνει το Συμβούλιο και η Κομισιόν, ειδικά στα ζητήματα της καθημερινότητας, ε, γιατί εδώ πέρα το Κοινοβούλιο έχει αποκτήσει περισσότερες αρμοδιότητες, αλλά ε, έχει δείξει κρίση πως σε τρεις σημαντικούς τομείς, δηλαδή κοινωνική πολιτική, οικονομική πολιτική και δημόσια οικονομικά, Ε, δεν υπάρχουν τα μέσα και συναπόφασης ε, και για να κινηθούμε με τρόπο συντονισμένο και αποφασιστικό. Αυτό το παρατήρησε ο πολίτης και αυτές τις αδυναμίες εκμεταλλεύονται αυτοί που θεωρούν πως η Ευρώπη είναι το πρόβλημα και όχι η λύση. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και η δική μας η αποστολή είναι νομίζω να ασκήσουμε πίεση να υπάρξει περισσότερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεύτερον να πείσουμε τους πολίτες πως η επιστροφή στον ε, εθνικισμό ή ε, στις περιφέρειες δεν μπορεί να είναι η απάντηση. Κύριε Γκερέρο Σαλόμ. Ευχαριστώ που ήρθατε να μας ακούσετε και να μας υποβάλλετε ερωτήσεις και να μας ζητήσετε τη γνώμη για ό,τι σας ενδιαφέρει. Και εγώ σαν καλός ευθύς και καλός ε, Ισπανός, δεν ξέρω ποιο προηγείται, ετοίμασα μια εισήγηση μισή ώρας για να σας εξηγήσω ποιο είναι το πρόγραμμα των σοσιαλδημοκρατών. Αλλά θα προσπαθήσω τελικά να σας τα πω περιληπτικά ακριβώς όπως ζητεί και η Προεδρεύουσα της Συνεδρίας της για τις Πρώτες Εκλογές οι οποίες θα γίνουν ε, μετά ή τέλος πάντων ε, την ώρα που σοβεί αυτή η τελο παντων την ωρα που κρίση και πρώτη για κάποιες εκλογές που σε αντίθεση με το παρελθόν μας δίνουν την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε δύο διαφορετικές συνταγές εξόδου από την κρίση. Διαφορετικά προγράμματα, προτάσεις διαφορετικές για το μέλλον. Τι λέμε οι σοσιαλιστές. Θέλουμε αλλαγή θέλουμε αλλαγή με τις εκλογές αυτές. Αλλαγή στην οικονομική, πολιτική αλλαγή, στη γενική ρότα που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εκλογές ούτως ώστε να διατρέψουμε τις πληγές αυτές που έγιναν βασικά στην κοινωνική πολιτική και όσον αφορά την κοινωνική συνένεση σε σχέση με το ευρωπαϊκό όραμα, δηλαδή με αυτές τις εκλογές θέλουμε να χτίσουμε να δημιουργήσουμε μία ισορροπημένη πρόταση για την Ευρώπη ούτως ώστε να ξεφύγουμε από αυτή τη μονοδιάστατη άποψη για την ε, οικονομική, ε, ε, οικονομική διαχείριση και διακυβέρνηση και μην έχουμε την παρεμβατική πολιτική Επομένως, Αλλαγή πρώτον. Δεύτερον, ε, να γιατρέψουμε τις πληγές και τρίτον, οικοδόμηση, δημιουργία. Οπότε και εμείς και αυτό κάνουμε γιατί αυτό προσδοκούν οι πολίτες και γι' αυτό θέλουμε να κατεβάσουμε ε, και έναν υποψήφιο για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε και την άλλη πολιτική ομάδα της, ε, του Κοινοβουλίου και δεν θα κατέβει σε εκλογές ο υποψήφιός τους και θα ήθελα ε, να πω, όπως είπε στο τέλος ο κ. ότι αν το κοινοβούλιο είναι αυτό το οποίο έχει την δημοκρατική το κοινοβούλιο, λόγω των αμέσων εκλογών, και αν κάποιος ε, θέλει να προεδρεύσει τις Κομισιόν ε, θα πρέπει να, να αναβαπτιστεί μέσω των εκλογών αυτών. Κλούτε. Σας ευχαριστώ, έρχομαι από τη Γερμανία. Επόμενος θα μιλήσω και γερμανικά. Υπάρχει γενικά συνένεση σε κάτι για το οποίο νομίζω και οι τρεις συμφωνούμε παρά το γεγονός ότι ερχόμαστε από διαφορετικά πολιτικά κόμματα ότι δεν πρέπει η Ευρώπη να αντιμετωπιστεί ως ε, πρόβλημα, αλλά ως η λύση που απαιτείται και ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε τις απαραίτητες λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν βέβαια διαφορές μεταξύ μας. Εγώ έρχομαι από ένα αριστερό πολιτικό κόμμα και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι μια δημοκρατία μπορεί να έχει πράγματι νομιμοποίηση μονάχα όταν εξασφαλίζει την ευμάρεια των πολιτών της. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν αρκεί να λέμε ότι η Ευρώπη είναι δημοκρατική όταν οι δημοκρατικές διαργασίες υπάρχουν, οι τυπικές διαδικασίες είναι δημοκρατικές και διαφανείς. Χρειαζόμαστε όμως και μια κοινωνική νομιμοποίηση η οποία προκύπτει μονάχα από την εξασφάλιση της ευμάρειας. Αυτό ήταν και μία από τις σημαντικές εμπειρίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι η δημοκρατία στην ε, Δυτική Ευρώπη ενισχύθηκε και εδρεώθηκε ακριβώς γιατί εξασφαλίστηκε ότι χάρη στο δημοκρατικό πολίτευμα μπόρεσαν να εξασφαλίσουν οι δυτικές κοινωνίες μια οικονομική ανάπτυξη στην οποία συμμετείχαν όλοι ή τουλάχιστον με ένα τέτοιο τρόπο συμμετείχαν ώστε να θεωρούν ότι υπήρχε κάποια δικαιοσύνη πίσω από αυτή την κατανομή του πλούτου. Η κρίση όμως ακριβώς είχε το αποτέλεσμα να αυξήσει τις ανισότητες στην Ευρώπη και να φέρει την Ευρώπη σε μια κατάσταση έλλειψης ισορροπίας. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, ιδίω στην Νότια Ευρώπη, που θεωρούν ότι αποκλείονται από την οικονομία και την κοινωνία λόγω της πολιτικής που ακολουθήθηκε από τις κυβερνήσεις τους, νιώθουν να είναι απόκληροι σε σχέση με την ευμάρεια και θεωρούν ότι αυτοί είναι τα θύματα ενός ε, συστήματος το οποίο έχει τις δικές του αδυναμίες, τις οποίες όμως πληρώνουν όχι οι ισχυροί και οι μεγάλοι, αλλά οι μικροί και οι φτωχοί. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Εάν δεν μπορέσουμε να επιλύσουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μακροχρόνιο δημοκρατικό πρόβλημα το οποίο θα προκύψει από αυτή την κατάσταση και την αντίληψη. Και δεύτερον, θέλω να, επι... να επαναλάβω ότι η Ευρώπη δεν είναι το αίτιο, δεν είναι το πρόβλημα είναι η λύση, γιατί η λύση μπορεί να προκύψει μονάχα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κρίση λοιπόν μας κατέδειξε ότι ο δρόμος της ε, ολοκλήρωσης που έγινε μέσα από το ευρώ και εγώ θεωρώ ότι το ευρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια οικονομική ολοκλήρωση. Η κρίση έδειξε ότι δεν μπορεί κανείς να έχει μια νομισματική ένωση με το ευρώ χωρίς να υπάρξει και, και ολοκλήρωση σε επίπεδο δημοσιονομικό και σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής. Δεν υπάρχει λοιπόν διαφωνία σε σχέση με το θέμα αυτό, αλλά το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτή την ολοκλήρωση. Υπάρχουν ιδέες σε σχέση με το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και άλλες προτάσεις και εκεί είναι διαφορετικές οι απόψεις που δίνονται από τα διάφορα πολιτικά κόμματα. Πιστεύω όμως ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε το στόχο της ευρύτερης ολοκλήρωσης σε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δύο ακόμα σχόλια πρέπει να κάνω. Από τη μία πλευρά φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά την ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πως μια, πως μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος, η Πορτογαλία, το Βέλγιο ή η Ελλάδα θα βρεθούν σε θέση να επιβάλλουν μια ρύθμιση των ε, αγορών αυτών. Ακόμα και η Γερμανία που είναι η πιο εύρωστη οικονομικά χώρα στην Ευρώπη δεν μπορεί να το πετύχει. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να επιτύχουμε μονάχα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να είναι τέτοιου χαρακτήρα ώστε να αντιλαμβάνονται και οι πολίτες ότι αυτό δεν είναι σε βάρος των απλών ανθρώπων ότι υπάρχει πράγματι μια αλληλεγγύη και δεν είναι προ όφελο μόνο των ισχυρών. Ένα δεύτερο σημαντικό ερώτημα είναι το θέμα του περιβάλλοντος, Τα πρόβλημα του περιβάλλοντο φυσικά δεν έχουν εθνικά όρια. Ξεπερνούν τα σύνορα, τα σύνορα είναι μια αφαίρεση μονάχα αλλά ο πλανήτης μας λειτουργεί σαν ένα σύνολο. Όλα τα οικολογικά προβλήματα λοιπόν ξεπερνούν τα στενά αυτά σύνορα. Αν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τα οικολογικά προβλήματα, θα είναι πολύ δύσκολο για τους πολίτες να καταλάβουν ποιο είναι το όνομα της Ευρώπης. Γι' αυτό χρειάζεται εμείς να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα ενισχύσουμε την ιδέα της Ευρώπης και να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι δεν πληρώνουν για να επωφεληθούν ορισμένοι μοναχά από τα χρήματα αυτά. Ωραία, κάποια ερωτήματα τώρα από το ακροατήριο, είτε για αυτά που είπε το πάνελ σας, είτε για τις εκλογές ε, του Μαΐου εν Παρακαλώ. Charles Fletcher από τα καλλιδονιακά μέσα στην Σκοτία. Όπως ξέρετε η Σκοτία έχει ένα δημοψήφισμα στις 18 Σεπτεμβρίου για την ανεξαρτησία της. Θα ήθελα να μου πείτε αν η Σκοτία πει ναι για να φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο, πόσο καλόδεκτη θα είναι στην Ευρωπαϊκή <clears throat> Ένωση ως 29ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως ο κύριος ισως ο κυριος κροσου Θα ήθελα να απαντήσω πάρα πολύ προσεκτικά γιατί τα ξέρω αυτά και από το Βέλγιο τις συζητήσεις αυτές. Και ως με ένας σχηματισμός 27 ε, χωρών ε, θα ήταν ε, πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε αύριο μια Ευρωπαϊκή Ένωση των 60-70 χωρών. Δεν ξέρω, θα πρέπει νομίζω ίσως να αναζητηθεί μια νέα μορφή συνεργασίας στο επίπεδο του Ηνωμένου Βασιλείου, μάλλον όχι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς θα απαντήσετε. Εάν ένας Βέλγος μας λέει ότι θα πρέπει να προσέξουμε, φανταστείτε τι θα σας πει ο Ισπανός. Νομίζω ότι τέτοιου είδου απαντήσεις που αρέσουν τόσο πολύ στους δημοσιογράφους. Ε, είναι, είναι πιασάρικες που λέμε, αλλά αυτά δεν βγαίνουν από τη συνθήκη. Δηλαδή δεν προκύπτει πιθανό ότι κάποιος βγαίνει από την Ένωση και δεν ανήκει πια εκεί και ε, δεν σημαίνει αυτό ότι κάποιος που βγαίνει δεν μπορεί να ξαναμπεί. Σημαίνει ότι δεν μπορεί ακριβώς θα θα βρεθεί στην ίδια χώρα, στην, στην ίδια θέση που βρίσκεται οποιαδήποτε τρίτη χώρα η οποία ζητεί την ένταξή της Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα γίνει έλεγχος όλων των ε, ε, συνθήκων, των προϋποθέσεων που πληρεί τυχόν αυτή η χώρα με τα κριτήρια της Κοπενχάγης, αν πληρούνται, ε, θα ελεγχθεί η συμβατότητα με το κοινοτικό κεκτημένο σε σχέση με την εθνική νομοθεσία αυτής της χώρας, αλλά πάνω απ' όλα πάνω απ' όλα, πάνω απ' θα πρέπει να υπάρχει ομοφωνία για την ένταξη στο Συμβούλιο. Γιατί αν δεν υπάρχει ομοφωνία στο Συμβούλιο δεν γίνεται η χώρα εκείνη η οποία προέκυψε από μια διάσπαση ενός κράτους μέλους να ενταχθεί ως μέλος στην Ένωση. Κλούτε. Κοιτάξτε, εγώ θα απαντήσω κάπως διαφορετικά μπορούμε να το δούμε ρεαλιστικά αν θέλετε οπότε έχουν δύο, οι δύο συναδελφοί δίκιο αλλά κοιτάξτε δεκαετία του 90 υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση για μια Ευρώπη των ε, περιφερειών και τότε το βλέπαμε ως μια ευκαιρία ότι δηλαδή αυτές οι περιφερειακές ε, σύγκρουσεις μπορούσαν να επιληθούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και αν θεωρούμε πως η Ευρώπη απομακρύνεται από τα εθνικά κράτη γιατί να μην συζητήσουμε αυτό το θέμα και να πούμε ναι μπορούμε να έχουμε και διαφορετικές περιφέρειες και δεν πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε τα εθνικά κράτη εντάξει εγώ είμαι κάπως ε, ριζοσπάστης δεν χρειάζονται θεωρώ εθνικά κράτη θα μπορούσαμε να έχουμε τα επίπεδα κάτω από το εθνικό κράτος και το ευρωπαϊκό επίπεδο, οπότε θα το λύναμε αλλιώς. Αλλά βεβαίως γνωρίζω πως είναι μια υπόθεση η οποία δεν θα λυθεί ε, φέτος, είναι κάτι το μακροπρόθεσμο. Οπότε θα μπορούσε, δεν ξέρω. Τι σημαίνει αυτό, θα έχουμε μια τεράστια κεντρική διοίκηση στις ε, Βρυξέλλες ή υπάρχουν κάποια επίπεδα διοίκηση στο πλαίσιο της επικουρικότητας ε, πιο κοντά στον ε, πολίτη. Ε, δεν θέλω κι εγώ ένα τεράστιο διοικητικό τέρας στις Βρυξέλλες αλλά θα ήθελα να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση και να ενθαρρύνω τους συναδελφούς με όλο τον ρεαλισμό που πρέπει να υπάρχει Νομίζω πως ε, με ευκαιρία την ε, Σκοτία μπορούμε να δούμε ε, πώς θα υπάρξει ένας δημοκρατισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα από τα εθνικά κράτη. Σας ευχαριστώ. Νομίζω πως θα εμπνεύσετε τους ακροατές μου. Ναι, ο κύριος εδώ. Τσίακμαν από την Λετωνία. Έχω ένα ερώτημα αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα εκλεγεί ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημαίνει πως θα έχει περισσότερες αρμοδιότητες ως εκτελεστική εξουσία σε σχέση με το νομοθετικό σώμα του Κοινοβούλου. Βλέπετε κάποια αναλογία δηλαδή με τα κράτη-μέλη. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι οι εκλογές παίρνουν τώρα και ένα πρόσωπο με τους επικεφαλείς των κομμάτων. Και επομένως θα πρέπει να έχουν κάποιες συγκεκριμένες γραμμές που παρουσιάζουν. Αυτό δεν ήταν πάντα έτσι. Είναι πιο εύκολο για τον κόσμο να καταλάβει ότι έχει το Juncker αντίον του Σούλτ παρά αφηρημένες γραμμές. Το θέμα όμως είναι ότι η Κομισιόν ε, ο, θα εκλεγεί ο πρόεδρος της Κομισιόν και η Κομισιόν θα πρέπει να σέβεται ορισμένους κανόνες. Είναι πολλά πράγματα όμως τα οποία δεν θα αλλάξουν. Δεν θα αλλάξουν οι αρμοδιότητες της Κομισιόν με αυτή την εκλογή. Είναι πιο σημαντικό να υπάρξει μια αλλαγή στην σχέση της Κομισιόν με το Κοινοβούλιο και κάνω εδώ ένα παραλληλισμό με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εγώ θεωρώ ότι πάντα ήταν ε, επικοδομητικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί δεν είναι απαραίτητο κάποιος να λέει πάντα ναι και ο άλλος να λέει πάντα όχι. Είναι λοιπόν πολύ πιο σημαντικά από το να διατηρηθεί μια πλειοψηφία όπως άλλα σε άλλα σε εθνικά κοινοβούλια. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα χάσει αυτή την ιδιαιτερότητα. Επομένως θα έχει το θάρρος να αλλάζει τις προτάσεις της Κομισιόν να τις απορρίπτει. Πιστεύω λοιπόν ότι αν γίνει απλώς μια διαμόρφωση κλίματος κυβέρνηση αντιπολίτευση αύριο θα χάσουμε πολλά πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι διαφωνώ με την πολιτική κατεύθυνση ότι αυτή τη στιγμή το μπαλάκι είναι στα χέρια του Συμβουλίου. Το Συμβουλίο δεν είναι αυτό το οποίο διορίζει τον πρόεδρο της Κομισιόν. Καθόλου. Το Συμβούλιο στέλνει ένα υποψήφιο για την προεδρία της Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν αυτό ο υποψήφιο, δεν αποσπάσει πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θα γίνει ποτέ πρόεδρος τη Επιτροπής. επομένω είναι απαραίτητο να συμπέσει η πολιτική γαλήνη από την πλευρά του Συμβουλίου, το οποίο δεν θα προσπαθήσει να κάνει παιχνίδια πολιτικάντικα σε αυτή τη διαδικασία και το οποίο θα στείλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως υποψήφιο για την προδία της Κομισιόν των επικεφαλής της πολιτικής ομάδας που έχει το μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι το άτομο αυτό θα γίνει πρόεδρος της Επιτροπής, γιατί θα πρέπει να έχει το ίμιση πλην πλέον ένα από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικοί συνασπισμοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να οδηγήσουν σε εκλογή ανθρώπων που δεν είναι κατά αναγκή επικεφαλής του πολιτικού κόμματος με τους περισσότερους βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά όλα αυτά σημαίνουν ότι οι πρόεδροι των τριών μεγάλων πολιτικών ομάδων, ο κύριος Ντόλο, ο κύριος Φερχόφστατ και ο κύριος Σφόμποντα, έχουν υπογράψει ένα κείμενο με το οποίο δεσμεύονται να ζητήσουν από το Συμβούλιο την μέρα μετά από τις εκλογές το Συμβούλιο να στείλει ως ε, υποψήφιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον επικεφαλής του κόμματος με τους περισσότερους βουλευτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει πρόεδρος, γιατί φυσικά απαιτείται πάντα η πλειοψηφία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις μια τέτοια αντιμετώπιση. Έχουμε τρία βασικά θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από αυτά τα τρία εκπροσωπεί άμεσα του πολίτε. Εκλέγεται άμεσα από του πολίτε. Ένα άλλο θεσμικό όργανο εκπροσωπεί τα συμφέροντα όλων βάσει της, ε, των ρητρών των συνθήκων, η Κομισιόν. Το τρίτο εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Έχουμε λοιπόν δύο δυνατότητες για το μέλλον. Είτε η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο που εκπροσωπούν με διαφορετικούς τρόπους το γενικό συμφέρον, το κοινό συμφέρον των πολιτών της Ευρώπης να δημιουργήσουν ένα συνασπισμό για να διαπραγματευτούν έναντι του Συμβουλίου. Αυτή είναι η θέση των σοσιαλιστών. Αυτό πρέπει να γίνει για μας. Ή αλλιώς ο πρόεδρος της Κομισιόν, που σας λέω και πάλι, στην, σε μια περίπτωση θα μπορούσε να μην είναι κάποιος στο παρελθόν που να εκτεθεί σε εκλογές, κάνει ένα συμβιβασμό με το Συμβούλιο, κάνει μια συμφωνία και κρατάει κοινή θέση με το, με το Συμβούλιο. Προφανώς λοιπόν υπάρχει αυτή η ανάγκη στην Ευρώπη να γίνονται διαπραγματεύσεις, να υπάρχει διαβούλευση και να υπάρχουν πολιτικοί συμβασμοί. Αλλά για μένα το σημαντικό είναι πώς θα υπάρξει η πολιτική πορεία στο μέλλον. Τα δύο θεσμικά όργανα τα οποία εκπροσωπούν το κοινό συμφέρον θα πρέπει να συνασπιστούν έναντι του Συμβουλίου που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των κρατών μελών σε εθνικό επίπεδο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να το τονίσω ακόμα περισσότερο έναντι της, ε, μέσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο κάθε αρχηγός κρατών και κυβερνήσεων βγάζει πάντα μια ανακοίνωση τύπου που να λέει πόσο κερδίσαμε εμείς και πόσα έχασαν οι άλλοι. Με αυτόν τον τρόπο όμως καταστρέφεται η Ευρώπη. Κοιτάξτε, και εγώ δεν θεωρώ πως οι αρμοδιότητες ε, θα αλλάξουν μέσω της άμεσης εκλογής του πρώτου Κομισιόν. Δεν, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στη συνθήκη, αλλά η πολιτική συμπεριφορά οπωσδήποτε ε, Κομισιόν και Κοινοβουλίου θα αλλάξει, κάτι το οποίο είναι σωστό και θετικό. Αν ε, οδηγήσει σε στενότερη συνεργασία, γιατί δεν είναι τόσο απλό πάντα απλή συνεργασία μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου. Αυτό εξαρτάται βεβαίω και από τον κάθε επίτροπο. Εγώ που δραστηριοποιούμε στα οικονομικά μπορώ να σα πω πως ο Μισελ Μπαρνιέ έχει πάρα πολύ καλή σχέση με την Επιτροπή μας, αλλά σε άλλους τομείς δεν ισχύει το ίδιο. Οπότε ελπίζω η σχέση Κομισιών και Κοινοβουλίου να βελτιωθεί. Οπότε θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γκρός ε, για τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου γιατί είναι δύσκολο να αντιληφθούμε την ε, διαφορά μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων γιατί πράγματι δεν υπάρχει συμπολίτευση και αντιπολίτευση που ένας λέει ναι και ο άλλος λέει όχι. Εδώ πέρα πραγματικά εργαζόμαστε πάνω στα ζητήματα και προσπαθούμε να διαμορφώσουμε κάποιες αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα δημοκρατικό έλλειμμα το οποίο υφίσταται βεβαίως θεωρητικά αλλά στην πράξη νομίζω πως είναι πιο ευρωπαϊκό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη Γερμανική Βουλή την οποία γνωρίζω ειδικά αν μιλήσουμε για συμμετοχή των ε, βουλευτών και δεν νομίζω πως το πρόβλημα είναι η σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν το πρόβλημα είναι μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ο ρόλος του Συμβουλίου είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξαναδούμε και εδώ πέρα η ε, επιθυμία μου είναι πραγματικά να μεταβληθεί η στάση του Συμβουλίου σε σχέση με τα όσα σχήνουν αυτή τη στιγμή. Όπως είπε ο κύριος ε, Σαλόμ, φαίνεται πως ε, η λιγότερο ευρωπαϊκή αντίληψη υπάρχει στο Συμβούλιο αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο το οποίο εμποδίζει τις ε, θετικές και τη θετική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ στο κέντρο της αιθούσης εσείς με το παλτό το κόκκινο. Ρώσο ονομάζομαι από την εφημερίδα Ελ τη της ε, Καταλανής. Δύο ερωτήσεις. Πρώτα πρώτα. Με την κρίση όλο ένα και περισσότερο είχαμε δυσπιστία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί είχαμε και τι φωτογραφίες, ε, ε, τις παλιές, τον κόλ με τον Μιτεράν που πήγαινε χέρι-χέρι. Αυτό ήταν μια φωτογραφία η οποία πια δεν πείθει τους νέους, τις καινούργιες γενιές. Αυτά όλα είναι τώρα προϊστορία. Δεν πείθαν τους νέους. Αλλά για πέστε μας, ε, ποια θα πρέπει να είναι η σημερινή μυθολογία ούτως υπήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να ξαναελκύσουμε τον κόσμο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να δει την πραγματική ε, υφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κόσμος. Επίσης κάτι άλλο. Άκουσα τι είπε ο κύριος Κλούτε. Μας μίλησε για τις σχέσεις Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου και Συμβουλίου από την άλλη μεριά. Τώρα πρόσφατα και ίσως και λόγω της κρίσης έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο έλλειμμα. Έλλειμμα δυσκολ... όσον αφορά τη δυσκολία δηλαδή της λήψης των αποφάσεων όποτε χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε δηλαδή για να πάρει και από αποφάσεις ο κ. Ντράγκη να σώσει το ευρώ, έπρεπε να γίνουν 15, μόνο 20 συναντήσεις κορυφής. Όμω θα έχουμε τώρα κάποιε μικρέ μεταβολέ στην Ευρώπη, μήπως ε, κάτι μπορεί να γίνει ούτω ώστε η Ευρώπη να μπορεί να λάβει κάποιες ε, ε, αποφάσεις πιο γρήγορα. Θα υπάρξει πιο ευέλικτη δυνατότητα λήψη αποφάσεων περισσότερο από ό,τι σήμερα. Πρόεδρος, να αρχίσουμε από εσά. Για πετε μας εσείς κύριε Γερέρο για την πρώτη ερώτηση για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, του ευρωπαϊκό όραμα. Η πρώτη ερώτηση αφορά αυτή την, την μυθολογία, αυτό το οποίο χρειάζονται οι νέες γενιές, ούτως ώστε να ε, θεωρούν ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι μέρος αυτού του οράματος το οποίο έχει μέλλον. Η δημοσιογράφος της εφημερίδας της Βαρκελόνης μας ε, ανέφερε εκείνη την εικόνα, τη φωτογραφία, την εικόνα ε, που, ήταν, είχε σημειολογική σπουδαιότητα του Νκόλ και του μητεραν χερι Έχουμε τον Φελίπε Γκονσάλες, τον Αντρεώτη επίσης, τον Ζακ Ντελόρ σε αντίστοιχες φωτογραφίες. Θέλω να πω ότι υπάρχει λόγος που υπήρχε αυτή η σημειολογία και στο μέλλον, επομένως αυτό που θέλουμε να υπάρχει ως μυθολογία είναι να μπορέσουμε να ανακτήσουμε ή πίν κάτι από την μυθολογία του παρελθόντος. Γιατί θυμάμαι ότι τέλος δεκαετίας του 80 ο Ζακ Ντελουτή έλεγε την Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγε ότι πρόκειται για μια ανταγωνιστική οικονομία. Αυτό είναι η Ευρώπη, έλεγε. Με ένα μοντέλο κοινωνικό και να υπάρχει και κάποια ε, εδαφική συνοχή και να έχει και αλληλεγγύη. Επίσης, στην ενακτήρια ομιλία του το 89, όταν ο Ντελόρ ανέλαβε τα ενία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τότε τι είπε σε αυτή του την πρώτη ομιλία, ότι χρειάζεται μια ψυχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ψυχή θα είναι η παιδεία, και ο πολιτισμός. Να, ο συνδυασμός αυτός που τώρα θα πρέπει να προσαρμοστεί στα του 21ου αιώνα. Αυτό χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται μια οικονομία ανταγωνιστική. Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια σκηνή. Ε, για να κοιτάξουμε ποιε είναι οι προοπτικές. Αυτές που χτες δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2015 θα δούμε ότι υστερούμε σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Άρα χρειάζεται το κοινωνικό μοντέλο να αναπτύσσεται χέρι-χέρι με την οικονομική διακυβέρνηση. Και για αυτό εμείς και οι σοσιαλιστές ε, ζητούμε ένα κοινωνικό σύμφωνο ε, προοδευτικό, το οποίο χέρι-χέρι να προχωρεί με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Και χρειαζόμαστε να υπάρχει συνοχή και συνέπεια εσωτερική στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχουμε ανισότητες μεταξύ Βορρά και Νότου σε σχέση με την εξωτερική κρίση. Χρειάζεται και αλληλεγγύη. Και γι' αυτό και αναφέρθηκαν αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα. Τα ευρωομόλογα, τις πολιτικές ε, ανάπτυξης, τις ε, κινήσεις της οικονομική πολιτικής που δημιουργούν ε, απασχόληση. Ένας στους τέσσερις νέους είναι άνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει ομένω αυτοί οι νέοι να δουν ένα νόημα σε αυτή τη μυθολογία του παρελθόντος. Ιδάλλως δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν υπάρχει αυτή η ικανότητα δυνατότητα να δοθεί ε, στους νέους να μπορούσαν να φτιάξουν τη ζωή τους. Και γι' αυτό σας περίπτωσα το τι έλεγε ο Ζακ Ντελόρ τότε είχε αναπτυχθεί λιγότερο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά νομίζω ότι θα, έτσι θα πρέπει να συγκρίνουμε την τότε Ευρώπη με την σημερινή. Αν μπορώ να συνεχίσω σε αυτό το σημείο για τους νέους που αναφέρατε. Έχουμε την πρωτοβουλία αυτή για την εγγύηση για τους νέους και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Έχουν εγκρίνει τέτοιες ε, πρωτοβουλίες. Ακόμα και από τον κύριο Τρισέ ακούγαμε καλά νέα για την οικονομία. Σε σχέση λοιπόν με την απήχηση που έχουν αυτές τις πρωτοβουλίες στους νέους. Πιστεύετε ότι όλε αυτέ οι πρωτοβουλίε θα φέρουν του νέου και πάλι στη δουλειά. Οι συνάδελφοί μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξέρουν τι συνέβη σε αυτήν τη θητεία με την εγγύηση για του νέους. Στο τέλο, η συμφωνία που επήλθε για τις, για τις προοπτικέ δημοσιονομικές προοπτικές ήταν η έγκριση ενός προγράμματος 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για 28 χώρες για 7 χρόνια αν κάνουμε τον υπολογισμό τώρα και λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό ότι η χώρα μου θα ήταν μία από τι χώρε που θα έπαιρνε τα μεγαλύτερα ποσά λόγω τη υψηλή ανεργία, αυτό θα σήμαινε ότι στην Ισπανία δεν θα ξεπερνούσαμε τα 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για την πρωτοβουλία αυτή της εγγύησης για τους νέους. Όταν έχουμε 3 εκατομμύρια νέους κάτω των 35 ετών που είναι άνεργοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Είναι φυστίκια, είναι πασατέμπος σε σχέση με το όγκο του προβλήματος. Εμείς έχουμε τονίσει, όχι μόνο οι σοσιαλιστές αλλά και άλλες ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πρόβλημα αυτό και λέμε στο εκλογικό μας πρόγραμμα ότι θα πρέπει να φτάσει τα 21 δισεκατομμύρια ευρώ η εγγύηση για τους νέους 3,5 φορέ το τωρινό ποσό λοιπόν, και αυτό δεν είναι κάτι που το βγάζουμε από ένα καπέλο, είναι η, αυτό το οποίο θεωρεί το Διεθνές, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας ως το ελάχιστο ποσό το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Θέλει κάποιο από εσά να επανέλθει για το θέμα αυτό. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ πως ε, συνολικά στα θέματα αυτά πρέπει να τονίσουμε την εταιρική σχέση μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην ε, βλέπουμε αυτό το οποίο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μία αντιπαράθεση κρατών και Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί το βλέπω τα τελευταία χρόνια βγαίνουν, βγαίνουν διάφοροι και λένε πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε το χ και το ψ σαν να ήταν κάτι ξένο προς εμάς η Ευρωπαϊκή Ένωση εγώ όπως σας είπα είμαι από μεθοριακή περιοχή και οι νέοι μας είναι δίγλωση και τρίγλωση και σε σύγκριση λοιπόν με τις γειτονικές μας περιφερειές έχουμε 5 με 6% λιγότερη ανεργία. Οπότε ε, όταν εγώ βλέπω το θέμα της ανεργίας των νέων σήμερα βλέπω πως είναι θέμα εκπαίδευσης γιατί κάποιες περιφέρειες είναι προσανατολισμένες σε παραδοσιακές ε, μεθόδους ε, αλλά βεβαίω εδώ πέρα δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, οικονομικά μπορώ να προτείνω κάποια κίνητρα. Πάλι και εδώ πέρα δεν έχει να κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί τα ποσά είναι περιορισμένα που έχει για μια τέτοια πολιτική αλλά αν υπάρχει η διάθεση για συνεργασία μπορούν να γίνουν ε, πολύ περισσότερα αλλά δεν μπορούμε να μετατοπίζουμε ε, συνεχώς την ευθύνη από το εθνικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί στο περιφερειακό. Οι νέοι λοιπόν στην ε, περιφέρεια μου θέλουν να μάθουν και στις δύο πλευρές των συνόρων θα, είναι οπωσδήποτε, θα έχουν οπωσδήποτε πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα και νομίζω αν απαντήσουμε σε αυτά τα ζητήματα έχουμε ήδη μία πρώτη απάντηση. Επίσης ε, το άλλο. Εγώ υπενθυμίζω στους ε, νέους ε, την ιστορία των Κόλ και Μητεράν ότι υπήρξαν πολιτικοί που δώσανε τα χέρια και αυτό δεν είναι ιστορία μόνο, είναι καθημερινή επικαιρότητα. Τα ζούμε αυτά τα πράγματα και υπάρχουν τομείς, πράγματι, μεταφορές, ενέργεια, όπου η συνεργασία στο ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη αύριο, γιατί αποτυγχάνει σήμερα, γιατί δεν υπάρχει η διάθεση, όπως είπα, διασυνοριακή συνεργασίας. Η ενέργεια είναι καλό παράδειγμα, οι μεταφορές επίσης. Ε, οι σιδηρόδρομοι αύριο, αύριο μπορεί να δημιουργήσουν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας εάν υπάρξει η θέληση να πάμε σε έναν ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο από τους εθνικούς. Για την Ισπανία ισχύει αυτό, την ε, Γερμανία, τη Γαλλία, την Πολωνία κτλ. Γιατί η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη και κολλάμε στο ότι δεν υπάρχει συνεργασία. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά ε, είναι κάτι νομίζω το οποίο μπορούμε να πούμε στους ε, νέους. Υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα. Υπάρχουν λοιπόν θετικά παραδείγματα, υπάρχουν ανάγκες σε κάποιους τομείς ε, που θα πρέπει να φύγουμε από τα εθνικά και περιφερειακά αντανακλαστικά. Και ίσως θα πρέπει και κάπου αλλού ε, κομισιόν ή κοινοβούλιο να αφήσουν κάποιες υποθέσεις να επιστρέψουν αυτές στις ε, περιφέρειες. Κύριε Κλούτε, σύντομα για τους νέους, αν θέλετε, αλλά και για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυσκίνητη όσον αφορά την λήψη αποφάσεων και χρειάζονται τόσο σύνοδοι κορυφής μέχρι να ληφθεί μια απόφαση. Ναι. Μπορώ να συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό με αυτά που είπε ο προλαλής σας. Η ειρήνη για την κεντρική Ευρώπη είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο εδώ και 60 χρόνια περίπου αλλά υπάρχουν πάντα απειλές όπως αυτή που βλέπουμε να υπάρχει στην Ουκρανία που θέτει ένα αμφιβόλο αυτή την κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το καταλάβουν οι νέοι. Είναι πολύ δύσκολο σε κάποιον που είναι 20 χρονών να του εξηγήσουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό της ειρήνης. Ακόμα και η δική μου η γενιά, εγώ γεννήθηκα το 1953, ακόμα και αυτή η γενιά δεν είναι εύκολο να κατανοήσει πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην Ουκρανία. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν πολύ περισσότερο για το σημείο αυτό. Όλα τα θέματα λοιπόν που έχουν να, πούνε με το, έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με την ενέργεια, με τις αλλαγές στον εργασιακό κόσμο, με την παγκοσμιοποίηση σε τελική ανάλυση, γιατί προσθέτω και τα θέματα του διαδικτύου. Όλα αυτά τα θέματα, όπως είπα στην αρχή της ομιλίας μου, αυτά είναι θέματα είναι θέματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα από μικρά κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τονίσουμε, να εξασφαλίσουμε ότι εκεί θα πρέπει να είμαστε πιστικοί προς τους νέους και οι νέοι μπορούν πράγματι να πιστούν. Αυτό έχει φανεί και με την εμπειρία που έχουν αποκομίσει οι νέοι με προγράμματα όπως το Εράσμους, ταξιδεύοντας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να πείσουμε τους νέους να μπορέσουν οι νέοι να έχουν μια καλύτερη αντίληψη για το γιατί κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίπεδο. Τα θέματα πολιτιστικά είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλους. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι πια ε, αυτονόητα. Θα πρέπει να ξαναφέρουμε όλα αυτά τα πράγματα στη συνείδηση των νέων, την ιστορία της Ευρώπης και αυτό είναι ένα θέμα και εκπαίδευσης και οι ίδιοι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι έχουν να κάνουν ένα σημαντικό να παίξουν σημαντικό ρόλο και οι δημοσιογράφοι ιδίω με τη δική τους δραστηριότητα θα πρέπει να φέρουν στο προσκήνιο τα ζητήματα αυτά. Έρχομαι τώρα στο άλλο ερώτημα <clears throat> για την ε, λήψη αποφάσεων. Το Συμβούλιο νομίζω ότι ο τρόπος που αντιμετώπισε την κρίση ήταν ε, λίγο καταστροφικός από πλευρά ταχύτητος λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει να βρούμε ταχύτερους τρόπους να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετώπισε νομοθετήματα όπως το Six-Pack, τα έξι νομοθετήματα που είχαν σε στόχο να δημιουργήσουν ένα άλλο μηχανισμό ο οποίος θα μπορεί να αντιμετωπίζει ταχύτερα τις κρίσεις. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα. Θα χρειαστούν δύο ή τρία χρόνια για να μπορέσουν αυτά να εφαρμοστούν και σε εθνικό επίπεδο Νομίζω ότι η γενική μας κατεύθυνση ήταν στο μέλλον <clears throat> θα πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις αντιμετώπισης της κρίσης με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς και πιο γρήγορες διαδικασίες. Και εγώ να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Ο... Είδαμε ότι υπάρχει σύγκληση των απόψεων στον την ενεργεία των νέων, γιατί από ό,τι είδαμε υπάρχουν πολλοί τρόποι με του οποίου δεν μπορούσε κανεί να, να, να δει τα πράγματα. Και έχουμε την κάθε πολιτική ομάδα που έχει το τη γιατί εμεί θέλουμε να υπάρχει κάποιο είδου επένδυση, κάποιο είδου πρόγραμμα, να μην υπάρχει μόνο λιτότητα σαν πολιτική. Και ένα από τα βασικά θέματα θα ήταν το να υπάρχουν επενδύσει στην παιδεία, στην ε, ενημέρωση, στην ε, ε, έρευνα, στην ανάπτυξη. Και υπάρχουν επίση και άλλα θέματα όπου συγκλίνουν όλε οι πολιτικέ ομάδε, δηλαδή η επένδυση στην παιδεία. Πρόκειται για ένα αίτημα ε, για κάτι το οποίο τώρα το προωθεί η γαλλική κυβέρνηση και θα μπορούσαμε να δούμε πέραν του, του, του, του προγράμματος για την εγγύηση για τους νέους να έχουμε και άλλο είδους δράσεις και έτσι αυτό να μπορούσε να είναι επιτέλους καλά μαντάτα για τους νέους. Εν κατακλείδη θέλω να σας πω ότι αυτό που θέλω να δοθεί μια απάντηση ευρωπαϊκή, να μην πέσουμε ξανά στην παγίδα του ότι ό,τι πάει καλό το έκανε η εθνική κυβέρνηση, κάθε εθνική κυβέρνηση και ό,τι πάει στραβά ε, είναι κάτι το οποίο το έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτή φταίει. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τις ε, δυνατότητες στις εθνικές κυβερνήσεις. Και έτσι θα πρέπει επομένως όλοι να αισθανόμαστε ότι εκεί ανήκουμε. Άλλε ερωτήσει, οι οποίε παρακαλώ να είναι συγκεκριμένε, να επιστρέφονται γύρω από το θέμα των εθνικών εκλογών. Εκεί, εκεί πίσω βλέπω κάποιον σηκώσει το χέρι, κάποιος από εδώ. Πρώτα πρώτα να σας πω για το τι αλλαγές θα γίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είπαμε ότι θα έχουμε περισσότερους βουλευτές από την ακραδεξιά, από την ακραριστερά, από τα κόμματα τα ευρωσκεπτικιστικά και έχουμε επίσης την επικεφαλής του Γαλλικού Front National η οποία λέει ότι πιστεύει ότι θα μπορέσει να είναι να φτιάξει πολιτική ομάδα με ευρωβουλευτές από παντού οι οποίοι να σημαίνουν τις απόψεις της. Εσείς κύριε κύριε Ρωσαλόμ, για πέστε μας. Πόσο διαφορετικό πιστεύω ότι θα είναι το επόμενο κοινοβούλιο Θεωρείτε ότι αυτές οι ανησυχίες του κόσμου ότι θα έχουμε πιο, πολλούς, ε, πιο πολλά ριζοσπαστικά στοιχεία, ότι αυτό θα ισχύσει. Σαλό, πρώτα πρώτα σας λέω ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές ε, θα είναι πάντοτε ε, οι πιο πικάντικες από αυτές που πάντοτε υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ευρώπη. Ε, γιατί είπαμε ότι έχουμε τις ε, δημοτικές εκλογές, τις ελληνικές εκλογές και τις ευρωπαϊκές. Ε, άλλα χαρακτηριστικά για διάφορους λόγους. αλλάζει η εκλογική περιφέρεια θα μπορούσαμε να πούμε σε κάποιες χώρες άλλες δεν υπάρχει εκλογικό μέτρο το κατόφλι ε, αλλού είναι θέμα η, η αποχή πόσο κόσμος κατέβει ψηφίσει πάντως αυτό το οποίο είναι σήμερα γεγονό είναι το εξή, να το πω έτσι αισιόδοξα. Δύο-τρία πράγματα που γνωρίζουμε. Πρώτα-πρώτα ότι θα έχουμε περισσότερου ε, που θα είναι προσκεπτικιστέ, εξτρεμιστέ κλπ. Αυτό είναι κακά μαντάτα. Το δεύτερο το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι το μέγεθος δεν θα είναι αρκετό ούτως ώστε να αλλάξει την ενεργή στο κοινοβούλιο, το μέγεθος εκείνων. Θα υπάρξουν αλλαγές για άλλους λόγους και όχι λόγω του μεγέθους αυτών των πολιτικών ομάδων ή τέλο πάντων του αριθμού τέτοιων βουλευτών ε, ε, ακραίων. Επίσης αυτοί οι εξτρεμιστές θα είναι και ο ε, αντίθετος από τον άλλο. Είμαι πολιτολόγος και ότι όλα αυτά τα σας τα λέω και από επαγγελματική παραμόρφωση. Δηλαδή, εμείς οι πολιτιολόγοι μιλούμε για μια διμερή, διμερή συνασπισμό ε, ή ένα διπολισμό. Έχουμε επομένως δεξιά και αριστερά, ε, οπότε δεν μπορούν να τα, βρουν οι δεξί και αριστερούς και το, το, το, κέντρο τα πάει καλύτερα. Επομένως θεωρώ ότι εδώ πέρα θα έχουμε τις, τις βασικές πολιτικές ομάδες. Ε, αυτοί, αυτοί θα τα πάνε καλύτερα. Εμείς οι τρεις που, είμαστε εδώ, φιλελεύθεροι, πράσινοι και εμείς και νομίζω ότι τελικά το, ο κίνδυνος δεν είναι στο πώς θα είναι εκείνοι οι βουλευτές. Το θέμα είναι το κατά πόσον μπορούν εκείνες, θα είναι εκείνες οι πολιτικές μας, εκείνοι οι βουλευτές με κάποιο είδους δυναμικές κοινοβουλευτικές να απευθυνθούν στον κόσμο και έτσι να μπορέσουν να διαμορφώσουν, να σημαδέψουν, να αμαυρώσουν τις ε, στρατηγικές των άλλων πιο μεγάλων πολιτικών ομάδων. Να, για να μην κατονομάσω κάποια χώρα. Ας φανταστούμε τη χώρα Χ, τη χώρα Α. Το σημαντικό δεν είναι τι θέση θα πάρει μια ακραία πολιτική ομάδα, αλλά τι θα γίνει με το εάν τα άλλα τα πιο μεγάλα κόμματα επηρεάζονται και διαμορφώνεται η πολιτική τους από αυτό το εξτρεμιστικό κόμμα. Καταλαβαίνετε, μπορούμε όλοι να σκεφτούμε ποια χώρα διατρέχει τώρα στην Ευρώπη αυτόν τον συγκεκριμένο κίνδυνο. Πρόεδρος, κύριε Κλούτε, να σας απευθύνω το ίδιο ερώτημα. Ας πούμε το UKIP στο Ηνωμένο Βασίλειο κερδίζει ένα σωρό έδρες, όπως λένε άλλωστε και τα Γκάλο. Έχουμε επίσης και το κόμμα της Μαρή Λεπέν, Είπαμε και εκεί, θα, τον δεν θα πάνε καλά και λένε ότι οι ευρωσκεπτικιστές θα κάνουν με τη Μαρή Λεπέν μια πολιτική ομάδα. Αλλά ας πούμε ότι θα έχουμε πολύ περισσότερου από το UKIP και πολύ περισσότερου ευρωβουλευτέ, από ριζοσπαστικά κόμματα, ακραία κόμματα στο επόμενο κοινοβούλιο. Ο κ. Γκερέρα λέει ότι αυτό δεν θα επηρεάσει ε, την πορεία του κοινοβουλίου. Αλλά εάν όλοι αυτοί όμω ε, ενωθούν δεν θα μπορέσουν να αλλάξουν την ρότα, την πορεία, να θέσω το πρόβλημα κάπως διαφορετικά. Είναι προφανώς διαφορετική κατάσταση η οποία θα προκύψει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Τα κόμματα αυτά τα οποία θα έρθουν ε, και θα είναι τη άκρα δεξιά, θα έρθουν κυρίως από την Βόρεια Ευρώπη στις χώρες της ε, Νότιας Ευρώπης δεν είναι τόσο έντονη η δύναμη των δεξιών κομμάτων. Οι χώρες λοιπόν αυτές που εξέθρεψαν σειρά δεξιά κόμματα είναι αυτές οι οποίες δεν έχουν φύγει ιδιαίτερα από την κρίση. Αυτή είναι η δική μου. από την Ελλάδα. Επομένως, η κατάσταση η οποία έχει προκύψει στις χώρες αυτές είναι ότι τα άτομα έχουν χάσει την ε, ευμάρεια που είχαν, έχουν χάσει τον πλούτο τους ως αποτέλεσμα της κρίσης. Επομένως υπήρξε μια αμυντική στάση στις χώρες του Νότου και τις χώρες της κρίσης, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαφορετική η στάση. Το UKIP έχει μια δική του άποψη για τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου προς την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δεν υπάρχει όμως το ίδιο πρόβλημα όπως αυτό της απώλειας αγοραστικής δύναμης και πλούτου όπως ε, στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Επομένως, το πραγματικό ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε εμείς να απομονώσουμε τις δυνάμεις αυτές. Εγώ φυσικά δεν είμαι κάποιος ο οποίος να υποστηρίζει αυτά τα δεξιά ριζοσπαστικά κόμματα. Έχω μια διαφορετική αντιμετώπιση για την ε, πολιτική. Το ερώτημα όμως πρέπει να θέσουμε είναι γιατί ο κόσμος έχει ριζοσπαστικοποιηθεί τόσο πολύ. Και αυτό δεν είναι θέμα μονάχα ισορροπίας δυνάμεων. Εδώ συμφωνώ με, τους, με τον Ισπανό συναδελφό μου. Τι γίνεται με τα άτομα τα οποία έχουν περιθωρικοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα, συγκεκριμένε ανησυχίε στα κρατη που βρίσκονται στην πηγή αυτού του φαινομένου. Αν δείτε τη ρητορική τη Μαρίν Λεπέ, είναι φορτωμένη με κοινωνικά θέματα. Είναι θέματα τα οποία δεν μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι απέχουν τόσο πολύ από διεκδικήσεις των αριστερών κομμάτων στην Ευρώπη. Λέει η Μαρίν Λεπέν ότι θα πρέπει να υπερασπιστούμε για την ε, ευμάρεια του μέσου εργάτη στην Γαλλία εναντίον στην Ευρώπη. Επομένως πρέπει να επανέλθουμε στην ε, αντιμετώπιση της ανησυχίας και των φόβων των ανθρώπων οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν μια πραγματική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά όλους αυτούς τους φόβους. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι με κάποιο τρόπο θα τους αποδιώξουμε, ότι αρκεί να έχουμε μια συγκεκριμένη ε, επιχειρηματολογία για να περιορίσουμε τα δεξιά κόμματα και τα ακραία κόμματα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά στη ρίζα τους, τους βασικούς αυτούς φόβους. Και εγώ. Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω καθόλου αυτές τις ε, τάσεις. Ε, και πρέπει να αναζητήσουμε κάποιες απαντήσεις γιατί το, το παιχνίδι το ξέρουμε οπωσδήποτε είναι πολύ πιο δύσκολο να είναι κανείς υπέρ της αλληλεγγύης αντί υπέρ του εγωισμού αλλά δεν είναι μόνο οι πλούσιοι που θέλουν να ε, αμφισβητήσουν την Ευρώπη. Βλέπετε πως ε, το εθνικό μέτωπο της ε, Γαλλίας ε, έχει, ε, ναι, έχει δύναμη σε κάποιες πλούσιες περιοχές αλλά και στην Μασαλία που έχει το που έχει άλλο πρόβλημα αυτό της μετανάστευσης οπότε το πρόβλημα είναι πρώτον η ανισότητα δεύτερον το πρόβλημα των αλλοδαπών ε, και βεβαίως ε, μια κάποια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αν δούμε την Ολλανδία, τη γειτονική μου χώρα, όπου τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολύ έντονη τάση τέτοια, αλλά η χώρα πραγματικά αυτή έχει κερδίσει πάρα πολύ από την Ευρώπη, γιατί είναι πολύ ισχυρότερη οικονομικά ε, από ό,τι ήταν πριν. Η τάση όμως είναι η τάση των πλουσίων αν θέλετε. Δηλαδή θα έχω μόνο τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης και τίποτα άλλο. Πρέπει να ξεχαρίσουμε στους ανθρώπους πως δεν υπάρχει μία ε, λύση που προτείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Καμία. Ε, έξοδος από το ευρώ δεν είναι λύση. Το πρόβλημα της μετανάστευσης ε, ήταν, είχαν την εξουσία σε κάποιες περιφέρειες, δεν ε, μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Και τέλος, επειδή ζω και στο Βελγίο, δεν είναι δυνατόν να μετατοπίζουμε την ευθύνη στους άλλους ε, κοιτάξτε, εμεί στο Βέλγιο έχουμε μια άλλη κατάσταση όπου δεν μπορεί ο καθένα να ψηφίσει όποιον θέλει, γιατί είναι στην ε, περιφέρειά του και έχει τα κόμματα τη περιφέρειά του. Εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω τον κύριο Φερχόφστατ. Οπότε θα, εγώ θα έπαιρνα στα σοβαρά αυτές τι τάσει, αλλά θα πρέπει να απαντήσουμε με τρόπο επικοδομητικό να πούμε ποια είναι η πραγματικότητα έχουμε εδώ πέρα ανθρώπου ε, που είναι παραδείγματο χάρη στην Επιτροπή Μεταφορών και 10 χρόνια δεν έχουν πει τίποτα. Ε, ας κάνουν και τίποτα εδώ πέρα, όχι μόνο να φωνάζουν στι ε, χώρε τους. Α γίνουμε λοιπόν, αν θέλετε, κάπως πιο λαϊκιστές, αν θέλετε αυτή τη λέξη, αλλά να δούμε ποιο αναζητεί λύσεις για τους ε, πολίτες. Δηλαδή να κάθεται κάποιο εδώ πέρα, να μην κάνει τίποτα, μάλλον και δεν θα κάνει και τίποτα για τους πολίτες αύριο. Μάλιστα, έχετε με ερωτήσεις, ο κύριος εδώ πέρα. Ναι, δουλεύει τώρα το μικρόφωνο. Θα λέγατε λοιπόν πως ε, η σύγκρουση στην Ουκρανία θα επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών ή τουλάχιστον την εκστρατεία. Και μετά στην ε, θεωρία ακροδεξιά και ριζοσπαστικά αριστερά κόμματα είναι πολύ διαφορετικά αλλά και τα δύο ε, δεν ασκούν κριτική στον ε, Πούτιν. Γιατί συμβαίνει αυτό κατά την άποψή σας. Μάλιστα, ευχαριστώ. για την Ουκρανία, κύριε Γκερέρο, θέλετε να απαντήσετε, θα επηρεάσει τις εκλογές. Γκερέρο. Νομίζω ότι σε κάποιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα γεγονότα στην Ουκρανία έχουν σαφή επιρροή γιατί πρόκειται για μια σύγκρουση που θέτει εν κινδύνο την ευρωπαϊκή ε, συνείδηση και άποψη ότι η ειρήνη είναι αυτονόητη, είναι εγγυημένη για πάντα και έτσι μπαίνει ένα τέρμα εις ε, την έννοια, την αντίληψη για το ποια είναι η γειτονιά μας, ποια είναι τα σύνορά μας ε, και επίσης ξεκινάει τώρα μια πολεμική σε σχέση με την ενέργεια, με την προμήθεια ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε και βεβαίω αυτό σημαίνει ότι κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωση, ε, αυτές που είναι πιο κοντά στην σύγκρουση, ε, θίγονται περισσότερο, ε, τι αφορά περισσότερο, όπω με τον ενεργειακό αφορά τη Γερμανία. Ε, η θέση της Ευρώπη στον κόσμο είναι κάτι που έχει να κάνει με την Γαλλία ή, την, ε, ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Και υπάρχουν και άλλες χώρες όπου δεν είναι τόσο σημαντική η επιρροή. Ας πούμε δεν θεωρώ ότι στην Ισπανία ή την η το ηνωμενο βασιλειο και υπαρχουν και άλλε χωρες οπου δεν ειναι τοσο σημαντικη η επιρροη α πουμε δεν θεωρω οτι στην ισπανια η την ιταλια ε, υπάρχουν κάποιες ε, συνέπειες. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει εκεί ανησυχία σε αυτέ τι χώρε. απλώς. Δεν βλέπω κάποιες συνέπειες από πλευράς εκλογική. Όμως νομίζω ότι για το σύνολο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης η σύγκρουση εκεί ε, αποτελεί ακόμα μία σκιά αμφιβολία που είπαμε και προηγουμένω. ότι δηλαδή δεν είμαστε πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο και ότι έτσι παραβλάβεται το κοινωνικό μας ε, μοντέλο. Και ε, αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε την αντιπαράθεση βορρά-νότου, αλλά επιπλέον τώρα ε, έχει πάψει να ισχύει η παλιά βεβαιότητα, η παλιά σιγουριά. Οπότε, βεβαίω και από πλευρά εκλογική ή προεκλογική θα υπάρχει μεγάλη επίδραση των γεγονότων αυτών. So we're just tackling the second part Δεύτερη ερώτηση για τα ριζοσπαστικά κόμματα και το ότι δεν ασκούν κριτική στον Πούτιν. Τώρα τα εσωτερικά, τα εσωτερικά των ριζοσπαστικότερων κομμάτων δεν τα ξέρω, αλλά συνολικά θεωρώ πως ε, η σύγκρουση αυτή ε, ανέδειξε πως κάποιες χώρες αντιλαμβάνονται διαφορετικά από εμάς την δημοκρατία. Δεύτερον, πως ε, μπορεί να γίνει μια διάκριση που του εάν μιλάει κανείς ομόφωνα ως αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης ή από υποχρέωση. Θεωρώ λοιπόν πως υπάρχουν σήμερα νέοι που θέτουν το ερώτημα του ποιο είναι το σύστημα που θέλω εγώ αύριο. Θα λειτουργεί με τον χ τρόπο ή τον ψ. Και μετά τίθεται και το ζήτημα ε, ισορροπίας μεταξύ κριτικής ε, ή κυρώσεων. Ε, εδώ πέρα δεν είναι ζήτημα νομίζω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε των κομμάτων αυτών. Εντάξει. Άλλα ερωτήματα. Μπορώ να πω κάτι, λέει ο κύριος ε, Σαλόμου. Να κάνω μια προσπάθεια να είμαι λίγο πιο ελαφρός αν θέλετε και να σας αφηγηθώ κάτι που ίσως ξέρουν κάποιοι από εσά. Είναι κάτι που συμβαίνει πολλές φορές στην, ε, στις Βρυξέλλες αλλά με το χιούμορ εκφράζει πάρα πολύ σαφώς τις ελλείψεις και τις αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι εδώ και κάποιες δεκαετίες ο Χένρι Κίσιγκερ είχε πει ότι, ότι όταν κάποιος θέλει να μιλήσει με την Ευρώπη δεν ξέρει τι αριθμό τηλεφώνου να πάρει. Αυτές τις στιγμές σε σχέση με τις διαφορετικές θέσει που υπάρχουν με την Ευρώπη λέει κανείς ότι αν πάρει κανείς τηλέφωνο την Ευρώπη Υπάρχει ένα ε, αυτόματο τηλεφωνητή που λέει για τη θέση τη Γερμανία πατήστε το 1, για την Αγγλία το 2, για την Ιταλία πατήστε το 3 και τα λοιπά. Είναι φανερό ότι αυτό είναι βέβαια αστείο, αλλά είναι ένα αστείο το οποίο έχει κάθε ε, νόημα γιατί αντανακλά μια πραγματικότητα. Ας σκεφτούμε ποια έχει σταθεί η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λιβύη, στη Συρία, στο Μαλί, σε όλες αυτές τις ε, σειράξεις που έπρεπε να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και όχι μονάχα στην περίπτωση της Ουκρανίας όπου και εκεί διαφοροποιείται η θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τη γεωγραφική του θέση, με βάση τα συμφέροντα και τις οικονομικές ή ενεργειακές τους ανάγκες κτλ. κτλ. Εντάξει. Άλλα ερωτήματα. Όχι. Αν μπορώ εγώ να θέσω ένα ερώτημα σε εσά, κύριε Κλούτε. Καλύπτω τα θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα τελευταία πια τέσσερα χρόνια νομίζω και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από τη συνθήκη Λισαβόνα έχει αποκομίσει πολύ περισσότερες εξουσίες. Βλέπετε ότι και οι βουλευτέ νιώθουν να έχουν μεγαλύτερε εξουσίε. Μετά όμω γυρίζω στη χώρα μου και εκπλήσωμαι η Ιρλανδία λόγω των οικονομικών προβλημάτων, λόγω του δημοψηφίσματος έχουμε υποχρεωθεί να ενδιαφερθούμε για τα ευρωπαϊκά θέματα και μπορείτε να πείτε ότι γενικά είναι καλά πληροφορημένη η Ιρλανδοί για τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά ο αριθμός των ατόμων που δεν ξέρουν τους βουλευτές τους, είχαμε 12 τώρα, θα έχουμε 11 μόναχα, αυτό με εκπλήττει κάθε φορά. Είναι άτομα τα οποία γενικά ενδιαφέρονται για τις ειδήσει, για την επικαιρότητα, παρακολουθούν τα νέα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμα τόση πολύ, τόσα χρόνια μετά από την ένταξη της Ιρλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που οι απλοί πολίτες δεν νιώθουν να τους εμπλέκει αυτό που γίνεται εδώ και δεν θεωρούν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το δικό τους κοινοβούλιο. Ναι. Και στη Γερμανία τα ίδια γίνονται. Ακόμα και ο Μάρτιν Σούλτς ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως υποψήφιος τώρα για την ε, Κομισιόν μπορεί να είναι πιο γνωστός από τους άλλους ε, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά στη Γερμανία δεν είναι περίπου κανένας γνωστός από τους ευρωβουλευτές. Η εντύπωσή μου λοιπόν είναι γιατί πιστεύουν στη Γερμανία ότι όλα αποφασίζονται στο Βερολίνο. Ενώ είναι γεγονός ότι 70 με 80% της νομοθεσίας που έρχεται στην Bundestag είναι μονάχα η εφαρμογή ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η ρητορική όμως σε πολιτικό επίπεδο είναι πάντα αυτή και ίδια και να κάνω τώρα και μία παρατήρηση για τα μέσα ενημέρωση. Και τα μέσα ενημέρωση παίζουν αυτό το παιχνίδι. Ό,τι αρνητικό έρχεται έρχεται από τι Βρυξέλλε και ό,τι θετικό έρχεται από το Βερολίνο. Αυτή είναι η εντύπωση που δημιουργείται. Όσο λοιπόν δεν αλλάξει αυτή η κατάσταση και δεν έχουμε και μια πιο ισοδίκαια και διάφανη παρουσίαση των γεγονότων, δεν ξέρω πώς θα αλλάξει αυτό αλλά κατά τα άλλα έχω την εντύπωση ότι χάρη στην κρίση τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια στη Γερμανία αναφέρθηκαν πολύ περισσότερα στα μέσα για την Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Από το 2010-2011 έχει αρχίσει στα μέσα ενημέρωσης να υπάρχει περισσότερη έμφαση στα ευρωπαϊκά θέματα. Και υπάρχουν και άλλες χώρες βέβαια που έχουν ίσως διαφορετική κατάσταση. Οι Πορτογάλοι συνάδελφοι μου λένε ότι μια φορά τη βδομάδα τους καλούν στην πορτογαλική τηλεόραση και έρχονται βουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες που βγαίνουν στα παράθυρα βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ζητάει κανείς να ε, δώσουν τη γνώμη τους για την οικονομική κρίση κτλ. Και στην Ελλάδα φαίνεται ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ίσως επειδή η Ελλάδα έχει πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση, υπάρχει μια μεγαλή, ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το τι γίνεται στις Βρυξέλλες, πώς αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντά μας οι ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες και τι κάνουν. Αλλά γενικά η κατάσταση νομίζω ότι είναι αρκετά πολύπλοκη και πολύμορφη. Απλώς θέλω να τονίσω ότι εμείς ως πολιτικοί εξαρτώμεθα από τη βοήθεια των δημοσιογράφων Γι' αυτό κάνω και αυτή την έκκληση προς εμάς με ύψιλον. Δεν θέλω να έχω αρνητική άποψη για τα μέσα ενημέρωσης, δεν θέλω να σας υποτιμήσω, αλλά θέλω να κάνω αυτή την έκκληση προς, ε, προς εσάς. Σας παρακαλώ χρησιμοποιήστε την ευκαιρία αυτή να λέτε περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και με διαφοροποιημένο τρόπο. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό για τους βουλευτές οι οποίοι είναι εδώ στις Φρυξέλλες, παραγωγός για τους γερμανούς δημοσιογράφους, να επιβάλλουν την άποψή τους σε ένα έντυπο που εκδίδεται στο Βερολίνο ή κάπου στη Γερμανία, αλλά είναι απαραίτητο τα μέσα ενημέρωσης να μετα... μετατρέψουν λιγάκι τη θέση τους και να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά θέματα. Υπήρξε η Press Europe στο Παρίσι, υπήρξαν πολλές ομάδες δημοσιογράφων που έχουν προσπαθήσει κάθε μέρα να δίδουν ε, ειδήσει για τα ευρωπαϊκά όργανα που μεταφράζονται σε διάφορες γλώσσες στα μέσα ενημέρωσης και ε, επομένως υπήρξε περισσότερο ενδιαφέρον για μας ως Ευρωβουλευτές. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να ενισχύσουμε τα μέσα ενημέρωσης εκεί που δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνο τους, να τους βοηθούμε με μεταφράσεις παραγματικά χάρη όταν δεν μπορούν να μεταφράσουν τέτοιες ε, τις ειδήσει οι οποίες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Είναι λοιπόν ένα κοινό καθήκον και για τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς και θα ήθελα να υπάρξει καλύτερη συνεργασία και να μην περιοριστεί αυτό μονάχα ε, σε επίπεδο των μεγάλων πολιτικών κομμάτων, να μπορούν όλες οι απόψεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αντανακλώνται στο, στα μέσα ενημέρωση. Και εγώ συμφωνώ, λέει ο Ρίκε Σαλόμ, στην θέση του κυρίου Κλούτε. Είναι απαραίτητο να υπάρξει κάποια υποστήριξη για την πλευρά των δημοσιογράφων για να μεταλαμβαδεύονται προς τους πολίτες οι θέσεις και οι συζητήσεις στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσουμε σε γενικό επίπεδο είναι ότι ενώ οι συγκεκριμένες πολιτικές που είναι όλο και πιο ευρωπαϊκές, οικονομική πολιτική, η πολιτική του περιβάλλοντος, η πολιτική καταναλωτών κτλ. Όλα αυτά μπορεί να είναι όλο και πιο ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Η πολιτική σε βασικό επίπεδο, η αντιπαράθεση των κομμάτων παραμένει να είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εθνική και μόνο. Και επειδή λοιπόν είναι σε εθνικό επίπεδο αυτή η αντιπαράθεση, τα μέσα ενημέρωση εστιάζουν περισσότερο στην πολιτική αντιπαράθεση που είναι εθνικού χαρακτήρα και όχι τόσο στι ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Ο κ. Γιούνκερ, υποψήφιο του ΕΛΚ, που είναι ένα άτομο το οποίο εγώ αναγνωρίζω σε ό,τι αφορά την ικανότητά του στο να εξηγούν με αποτελεσματικό τρόπο τα προβλήματα και τις δυσκολίες, είναι ένα άτομο το οποίο είπε ότι ξέρουμε να κερδίσουμε τις εκλογές, δεν ξέρουμε τι κάνουμε μετά όμως αν κερδίσουμε τις εκλογές. Όλοι οι αρχηγοί κομμάτων λοιπόν και οι ηγέτες σε εθνικό επίπεδο σκέφτονται πάντα με όρους πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό αρέσει πάρα πολύ στα μέσα ενημέρωσης. Οι δημοσιογράφοι εδώ από την Ισπανία ξέρουν ότι ένα μήνα μετά από κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει η χώρα μία συζήτηση στα ισπανικά κόρτες. Ενώ στη Γερμανία γίνεται ένα μήνα πριν. Ίσως μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Γίνονται πέντε ώρες συζήτησης για το θέμα αυτό και στη συνέχεια είναι, υπάρχει ο χρόνος ε, ερωτήσεων, ερωτήσεις προς τον ε, αρχηγό της κυβέρνησης. Δυόμιση λεπτά κάθε μπορεί να κρατήσει 25-30 λεπτά και αυτό καλύπτει τα 90% των ειδήσεων που βγαίνουν από τους δημοσιογράφους στην ε, επικαιρότητα. Λοιπόν, πρέπει όλοι τα μέσα ενημέρωσης, όλοι αυτοί οι οποίοι ε, ενδιαφέρονται για την Ευρώπη να κατανοήσουν την ανισότητα η οποία υπάρχει πολλές φορές. Υπάρχει αυτή η ανισότητα η οποία δημιουργεί πολλά προβλήματα για τους πολίτες μας, διατρέφει, εκτρέφει μάλλον τα ακραία τα, τα ριζοσπαστικά κινήματα εγώ είχα δει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο CNN της Κριστιάνα Αμαμπούρ με την Κριστιαν Λαγκάρτ για τα θέματα της ανισότητας, όχι για το Δουνουτού, όχι για τις προοπτικές ανάπτυξης, μόνο για την κοινωνική ανισότητα. 25 λεπτά συνέντευξης με την Κριστιαν Αμαμπούρ. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θετικό και αν επαναληφθεί και αλλού θα έχει πολύ θετικό αντίκτυπο. Ναι. Μπορώ να συμφωνήσω πολλά από αυτά τα οποία ε, υπόθηκαν, αλλά πρέπει να πω πως δεν χρειάζεται ε, πάντα να ερχόμαστε ή να κουβαλάμε κόσμο στις ε, Βρυξέλλες. Καλό είναι να γίνεται και καμία συζήτηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στο Κοινοβούλιο. Εγώ θεωρώ πως οι επίτροποι μας επίσης πρέπει να πάνε στα εθνικά κοινοβούλια, αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη εδώ πέρα, να πάνε εκεί να συζητήσουν με τους υπεύθυνου. Αυτό έχει δύο πλεονεκτήματα. Πρώτον θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον για τον τύπο, μα αυτό να γράψουν μια έκθεση, και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την ε, Κομισιόν να πάνε να εξηγηθούν στους βουλευτές στα Εθνικά Κοινοβούλια. Αν υπάρξει αυτή η γέφυρα μεταξύ ε, Εθνικού και Ευρωπαϊκού ή αν δεν γίνει ε, μάλλον δεν θα έχουμε επικοινωνία με τους πολίτες. Γιατί βλέπουμε πως υπάρχει η δυνατότητα αλλά δεν χρησιμοποιείται. Νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η γέφυρα. Τον Μάρτιν Σούλτ, τον οποίο εκτιμώ, του είχα πει «Εντάξει, φέρτε ανθρώπους εδώ πέρα, αλλά πρέπει να στείλουμε και κόσμο στις χώρες να πάνε οι επίτροποι να